Bien, la séance euh, Συνεχίζουμε την ε, συνεδρίασή μας. Θα ήθελα να ζητήσω από όλους όσους δεν θα παρευρεθούν, κυρίως απευθύνομαι στους δημοσιογράφους, είτε να ε, αποχωρήσουν είτε να παραμείνουν. Ε, μην διαταράσσετε όμως τη διεξαγωγή των εργασιών μας. Είναι πολύ φορτωμένο το απόγευμα. Και θα μας απασχολήσει η ακρόαση ε, εκπροσώπων τεσσάρων πολυεθνικών εταιριών, δύο πάνελ, ένα ψηφιακό ας το πω έτσι με την Apple και την Google και ένα βιομηχανικό με τους εκπροσώπους ε, της εταιρείας IKEA και McDonald's. Ε, καλωσορίζω τους εκπροσώπους των επιχειρήσεων αυτών. Θα ήθελα να παρακαλέσω για το χρόνο αγόρευσης ε, να είμαστε ιδιαίτερα πειθαρχημένοι, διότι έχουμε πάρα πολλούς ε, καταγεγραμμένους ε, ομιλητές. Εξυπακούεται ότι θα υπάρξει πλήθος ερωτημάτων προς τους τεσσάρους εκπροσώπους, ταυτόχρονα σε 3,5 ώρες δεν θα μπορέσουμε να εξαντλήσουμε κάθε πτυχή, κάθε λεπτομέρεια των ερευνών που θέλουμε να διεξάγουμε για αυτές τις εταιρείες. Δεν μπορούμε ε, λόγω χρονοδιαγράμματος ε, παρά να ακούσουμε ε, τον ένα εκπρόσωπο μετά τον άλλον όμως δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να πάρετε χρόνο ομιλίας από την επόμενη εταιρεία. Και ο Ρολάν Γκρά θα κάνει τον αστυνομικό γιατί το ίδιο ισχύει και για τους βουλευτές τα μέλη της Επιτροπής. Οπότε θα, προ... θα κινηθούμε ως εξής. Όπως και μέχρι στιγμής θα ζητήσουμε στους συγκεκριμένους να κάνουμε μια πεντάλεπτη εισαγωγική παρουσίαση, μετά ερωταπαντήσεις, Q&A και κάθε ομιλητής παρακαλείται να απευθύνει το ερώτημά του σε μία ή και στις δύο εταιρείες, να το διευκρινίζουμε εδώ που παίρνει το λόγο. Εάν είναι και για τις δύο, έχουμε ένα χαρακτηριστικό πεντάλεπτο. Μια, σε μία, μια με την παραδοσιακή πεντάλεπτη ε, χρονοθυρίδα. Ε, αλλιώς θα έχουμε δύο διαφορετικές ε, τρίλεπτες, ε, αν είναι για τις δύο εταιρείε. Ε, τρία και δύο για την απάντηση δηλαδή. Ως συνήθως. Ένα και δύο. Τρία δηλαδή, ένα και δύο. Για την, ε, ένα για την ερώτηση, δύο για την απάντηση. θα ακούσουμε τους εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων και φυσικά θα έχουν ίσο χρόνο οι προσκεκλημένες για να απαντήσουν. Λοιπόν, υπενθυμίζω πως ε, η Επιτροπή ε, στην οποία είσαστε σήμερα και ε, αναμεταδίδεται ζωντανά στο διαδίκτυο η συνεδρίαση να το θυμίσω είναι δημόσιες εργασίες της Επιτροπής ε, σχετίζονται με τον εταιρικό ε, φόρο δε στο, τις πρακτικές δηλαδή που διαπιστώνται στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μετά τα όσα διαμήφθησαν πέρυσι σε παγκόσμιο επίπεδο συγκεκριμένα στον ΟΣΑ αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση στα θεσμικά όργανα της και σε σχέση με τις πρώτες αποφάσεις που λήφθησαν ε, για τις ε, αυτόματες ανταλλαγές πληροφοριών για τα tax ruling, για τις φορολογικές δηλαδή συμφωνίες των κρατών μελών και επί τη βάση μιας πρώτης σειράς συστάσεων της ειδική Επιτροπής που εκπονήθηκαν πέρυσι και επί τη βάση του σχεδίου νομοθεσίας που κατέθεσε ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιανουάριο θα μας ενδιέφερε να γνωρίζουμε πώς τοποθετούνται οι εταιρείες σας σε αυτό το ευρωπαϊκό αλλά και παγκόσμιο φορολογικό περιβάλλον εν εξελίξη Οι περισσότεροι έχετε αντιμετωπίσει δυσκολίε σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή και με κάποια κράτη-μέλη. Γνωρίζουμε ακροάσεις όπως αυτές που έχουν γίνει ε, στη ΣΥΠΑ, στην Αιγερουσία ή στη Βουλή την, ε, ε, την Αγγλική και θέλουμε να καταθέσετε τη μαρτυρία σας σε αυτά τα πλαίσια που προσδιορίσα. Μόλις. Θέλω να δώσω το λόγο την εκπρόσωπο της Apple, Κάθη Κέρνη ή και Τζούλια Μακρέι για πέντε λεπτά. Καλό απόγευμα κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Λέγομαι ε, Κάθη Κάρνη, είμαι αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Επιχειρησιακού Σκέλους της Apple ε, και εργάζομαι στο Κόρκ στην Ιρλανδία, στα κεντρικά γραφεία και είναι μαζί μου σήμερα η Τζούλια Μακρέι η οποία είναι υπεύθυνη για τα φορολογικά της Apple στην Ευρώπη και ε, έχει τη βάση της στο Λονδίνο. Ε, πρώτα απ' όλα σας ευχαριστούμε που μας ε, καλέσατε σε αυτή την ακρόαση. Η ε, φορολογική πολιτική θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να προωθήσει την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Η φορολογική μεταρρύθμιση είναι αυτή η οποία μπορεί να... η οποία ενδιαφέρει, είναι μια διαδικασία η ενδιαφέρει όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Ε, η Apple εδώ και πάρα πολύ καιρό έχει ζητήσει μεγάλες φορολογικές ε, μεταρρυθμίσεις έτσι ώστε να υπάρξει αύξηση των αγωνισμού, συνοχή των φορολογικών καθεστώτων και οικονομική ανάπτυξη. Η άποψή μας ε, όσον αφορά τις φορολογικές μεταρρυθμίσεις είναι σαφής και είναι πάντα σύμφωνα με το μότο της Apple, δηλαδή καλύτερα απλά παρά περίπλοκα. Πρέπει να είναι σαφής η φορολογική νόμοι και θα πρέπει να, έχουν, να παρουσιάσουν μεγάλη συνοχή. Η, η ασφάλεια δικαίου και η ποιότητα των, ε, της, ε, του εργατικού δυναμικού ε, είναι αυτά τα οποία οδήγησαν την Apple να έρθει στην Ευρώπη 36 χρόνια πριν. Ο Steve Jobs ξεκίνησε την Apple το 1976 και αμέσως κατάλαβε ότι θα έπρεπε να έχει και ένα σκέλος στην Ευρώπη και επέλεξε λοιπόν την Ιρλανδία ως κέντρο κατασκευής και διανομής. Στη δεκαετία του 90 η Apple ε, είχε πολλές ε, απώλειες ε, και άρχισε η μετοχή της να πέφτει σε ολόκληρο τον κόσμο. Παρά τους δύσκολους καιρούς, η Apple δεσμεύτηκε ότι θα ήθελε να κρατήσει αυτήν την βάση στην Ευρώπη και σήμερα είμαστε ιδιαίτερος περήφανοι γιατί έχουμε συμβάλει στη δημιουργία πολλών θέσεων εργασίας. Ε, και ε, ε, μέσω και των Apple Stores που δημιουργήθηκαν 8 χρόνια πριν δημιουργήσαμε ακόμα περισσότερες θέσεις εργασίας. Εμείς θεωρούμε ότι μέσα και από νέες εταιρείες και βιώσιμες όμως εταιρείες δημιουργήσαμε καλές θέσεις εργασίας ύψους ενός εκατομμυρίου αυτή τη στιγμή. Και πρέπει να σας πω επίσης ότι τον προηγούμενο χρόνο δώσαμε πάνω πάνω από 11 δις ευρώ για ε, να συνεργαστούμε με περισσότερους από 4.500 προμηθευτές, πολλοί εκ των οποίων ήταν μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό ε, σημαίνει ότι στηρίζουμε πάνω από 240.000 θέσεις εργασίας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ε, προβλέπουμε να επενδύσουμε ακόμα 1,7 δις ευρώ έτσι ώστε να δημιουργήσουμε νέα κέντρα δεδομένων στην Ιρλανδία και στην Δανία. Στην Ιρλανδία άμεσα απασχολούμε 5.500 ανθρώπους ανθρώπους, ε, δηλαδή 25% περισσότερους από το 2015. 93% των ε, των εργαζομένων μας στην Ιρλανδία είναι ε, πολίτες των, της, των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 44% δεν είναι υπήκοοι της Ιρλανδίας. Αυτό είναι κάτι για το οποίο πραγματικά είμαστε εξαιρετικά περήφανοι Επίσης, ε, ε, στο σύνολο των επιχειρηματικών μας ε, διαδικασιών στην Ιρλανδία εμπλέκουμε 18.000 ε, Θέσει εργασίας και 200 εκατομμύρια ευρώ. Ε, η Apple αυτή τη στιγμή είναι ο μεγαλύτερος ιδιωτικός ε, φορέας απασχόλησης στο Κόρκ και πρέπει να σας πω ότι πλέον θεωρούμε ότι από τη στιγμή που είμαστε συνεπείς έχουμε, έχουμε γίνει, η Apple δηλαδή έχει γίνει ο μεγαλύτερος καταβολέας φόρων σε όλο τον κόσμο. Πληρώνουμε φόρους όπου οπουδήποτε ε, λειτουργούμε και είμαστε ε, παρόντες επιχειρησιακά σύμφωνα ε, με τον νόμο. Στην Ευρώπη οι φόροι μας αντικατοπτρίζουν τις πραγματικές μας εργασίες και επιχειρήσεις σύμφωνα με την κατασκευή, την κατανομή και τις πωλήσει. Πληρώνουμε πάρα, πολλά, πάρα πολύ ψηλά ποσά επίσης στις ΗΠΑ Πολιτείες όπου 70.000 άνθρωποι εργάζονται στις επιχειρήσεις μας. Κάνουμε, συμμετέχουμε σε ε, πολυμερείς ε, συμφωνίες όπως η BEPS ας πούμε έτσι ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε με συνολικό τρόπο να συμβάλλουμε στην βελτίωση του φορολογικού ε, περιβάλλοντος. Θέλουμε και περιμένουμε να υπάρξουν συγκεκριμένες προτάσεις οι οποίες θα οδηγήσουν σε μια σωστή φορολογική μεταρρύθμιση η οποία θα βοηθήσει όλους μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κυρία μου λέει ο Πρόεδρος. Μιλή μιλήσατε 4 λεπτά και 59 δευτερόλεπτα, άρα δώσατε ένα δευτερόλεπτο από το χρόνο σας στην ε, ε, επόμενη ομιλήτρια. Στον ομιλητή από την Google. Ε, κύριε Πρόεδρε και μέλη της Επιτροπής, σας ευχαριστώ που με καλέσατε να βρίσκομαι ενώπιόν σας εισαγωγικά ηγούμε ε, των οικονομικών θεμάτων για Ευρώπη, ε, Μέση Ανατολή και Αφρική για την Google και έχω και τη φορολογική πολιτική και τα τελευταία έτη συμμετείχα σε συζητήσεις με τον ΟΣΑ, με θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εθνικές κυβερνήσεις και διάφορους βιομηχανικούς ομίλους. Παρακολουθώ και τις εργασίες δικές σας με ενδιαφέρον. Ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση συζητείται ε, και στις πολιτείες όλο και πιο έντονα και αλλού ε, η φορολόγηση των επιχειρήσεων. Δύο χρόνια ο ΣΑ έκανε μελέτες και πολλά κράτη-μέλη θέλουν τώρα να αλλάξουν την πολιτική τους και τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Google από την πλευρά της εδώ και καιρό ζητάει ένα σύστημα διεθνές, πιο συνεπές, πιο συνεκτικό και πιο απλό Χιλιάδε σελίδε είναι πολλές φορές η φορολογική νομοθεσία στα κράτη-μέλη και ε, ανησυχούν βέβαια για τη διάβρωση τη φορολογική βάση, αλλά υπάρχουν αλλού φορολογικά κίνητρα ελαφρύνσεις, ε, χαμηλός ε, ε, φόρος για τις επιχειρήσεις και επιστώσεις ευνοϊκές για την έρευνα και την κοινοτομία. Υπάρχουν σαφείς κανόνες και χρειάζεται πιο ε, στενός ε, διεθνής συντονισμός. Εμείς υποστηρίζουμε την πολύ πλευρή υποστήριξη από την G20, Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΩΣΑ, αλλά να μην είναι κουρελού το σύστημα. Ε, υπάρχει κίνδυνος διπλής φορολόγησης, ε, παρατεταμένης διενέξεις μεταξύ διαφόρων δικαιοδοξιών κτλ. Όπως ε, εξήγησε τον Νοέμβριο συνάδελφος Νίκ ε, ε οι κυβερνήσεις πρέπει να γράφουν τους κανόνες και επιχειρήσεις να τους στηρούν. Η Google είναι νομοταγής και ακολουθεί και τα φορολογικά και τα κίνητρα και τις υποχρεώσεις. Όχι μόνο εμείς χρησιμοποιούμε τις ευνοϊκές ρυθμίσεις που είναι γνωστές, ε, ευρέως ε, ε, προσβάσιμες και που χρησιμοποιούν σχεδόν όλες οι πολυεθνικές εταιρείες. Και όσο αλλάζουν οι κανόνες θα συνεχίσουμε να τους στηρούμε. Η Google είναι μια εταιρεία πολυεθνική, παγκόσμια, αλλά έχει τις περισσότερες επαφές στις Ηνωμένες Πολιτείες και πληρώνει τους περισσότερους φόρους. γιατί είναι τέτοιο το αμερικανικό σύστημα ε, όπου 3,3 ε, ε, δις πληρώσαμε πέρυσι και 80% στις Ηνωμένε Πολιτείε, γιατί εκεί φορολογούν και τον κίνδυνο και το τόπο που παράγεται το κέρδος. 19% ήταν η αύξηση και είναι περίπου αντίστοιχο ο συντελεστής ε, με τον Ευρωπαϊκό. Έχουμε γραφεία σε 40 και πλέον χώρες, εδρεύουμε στην Ευρώπη, στην Ιρλανδία με 5.000 υπαλλήλου που εξυπηρετούν την Ευρώπη, την ε, ε, Αφρική και τη Μέση Ανατολή. Παγκοσμίω έχουμε μάλλον στην Ευρωπαϊκή Ένωση 14.000 υπαλλήλου και έχουμε δισεκατομμύρια επενδύσεων σε εταιρικέ σχέσεις. Για να δούμε την κλίμακα λίγο όμως και τη σύγκριση έχουμε πάνω από 20.000 μηχανικού στι ΗΠΑ που σχεδιάζουν και παράγουν προϊόντα και υπηρεσίες. Και ε, σε αντίθεση με αυτό η μηχανική μα στην Ευρώπη είναι μόλι 2.000. Ε, συνεχίζεται η συζήτηση κατά πόσο ε, η φορολόγηση του εταιρικού κέρδους θα πρέπει να γίνεται διαφορετική. Ιδιαίτερα όταν υπάρχει μετατόπιση από τον τόπο που παράγεται το προϊόν και η υπηρεσία στον τόπο που καταναλώνεται. Αυτό θα πρέπει να το αποφασίζουν οι κυβερνήσεις. Οποιαδήποτε αλλαγή θα πρέπει να βασίζεται σε ευρεία συνένεση έτσι ώστε εταιρείε και οι πολίτες να έχουν εμπιστοσύνη στο παγκόσμιο φορολογικό σύστημα. Ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο στον εισηγητή μας, τον κύριο Κόφουτ. Παρακαλώ. Ε, Θέλετε να απευθύνετε τα ερωτήματά σε εμείς και στις εταιρείε. Ευχαριστώ. Μόνο για την Google ήθελα να ρωτήσω κάτι προς το παρόν, γιατί ξέρω ότι οι υπόλοιποι θα ρωτήσουν την εκπρόσωπο της Apple. Οπότε καλύτερα να, για, χρηστή διαχείριση του χρόνου να υποβάλω το ερώτημα σε μια εταιρεία. Ευχαριστούμε πάντως που ήρθατε. Και ήθελα να πω πως είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας διότι ε, εξετάζουμε το θέμα των παράνομων κρατικών επιδοτήσεων και των φορολογικών συμφωνιών που οδηγούν σε ε, ε, αθέμητους όρους ανταγωνισμού και αυτό είναι προνομιακό φυσικά για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και οι μικρομεσαίες πληρώνουν 30% περισσότερους φόρους. Κάτι δεν πάει καλά. Και οι πολίτες βλέπουν ότι διαβρώνεται η βάση για τον εταιρικό φόρο, είναι πρόβλημα αυτό. Βλέπουμε ότι τα φορολογικά έσοδα μεταβιβάζονται σε δικαιοδοτικές επικράτειες όπου δεν υπάρχει κανένας συντελεστής εταιρικού φόρου. Λοιπόν, ε, θα πρέπει να κινηθείτε κι εσείς προς τη σωστή κατεύθυνση. Ε, υπάρχουν γνωστές φορολογικές πρακτικές για την Google και δεν είσαστε και οι μόνοι, ήθιστε στις πολυεθνικές. Θα γίνω πιο συγκεκριμένο τώρα. Ε, κάποιες από τις, ε, κάποια από τα υποκαταστήματά σας ε, πληρώνουν royalties ε, σε μια οντότητα στις ε, Βερμούδες και έτσι έχουμε το γνωστό σύστημα double Irish και double Dutch δύο διαφορετικά συστήματα Αναγνωρίζετε ότι χρησιμοποιείτε αυτούς τους φορολογικούς παραδείσους για να φοροδιαφύγετε και μπορείτε να μας εξηγήσετε γιατί έχει την έδρα της η Βερμούδα η, εταιρεία στην οποία πληρώνετε εσείς ρόγελτης και γιατί συγκεκριμένα σε αυτό το νησί και όχι αλλού. Ευχαριστούμε ο Διευθυντής. Ε, ε, ευχαριστώ για την ερώτηση. Είναι καλή ευκαιρία για να διευκρινίσω κάτι. Για την φορολογική δομή στη Βερμούδα, Δεν ε, σχετίζεται αυτό με το φόρο που πληρώνουμε σε ευρωπαϊκές χώρες. Ε, διότι έχουμε τον συγκεκριμένο αριθμό υπαλλήλων, συγκεκριμένο αριθμό δραστηριοτήτων σε αυτές τις δικαιωτικές επικράτειες και ούτως ή άλλως οι υπολογισμοί θα ήταν οι ίδιοι με ή χωρίς αυτή την οντότητα. Γιατί υπάρχει όμως, διότι υπάρχει μια ιδιαιτερότητα στο φορολογικό σύστημα των ΗΠΑ, ε, δηλαδή σε παγκόσμια και όχι σε εδαφική βάση υπολογίζεται ο φόρος ε, αντίθετα με τις ευρωπαϊκές χώρες και επειδή ε, ε, η ε, IRS, η αρμόδια αρχή των ΗΠΑ, διαρκώς ελέγχει τις ροές χρημάτων, θα πρέπει να ξεκαθαρίσω ότι μεταφέρονται οι φορολογικές υποχρεώσεις και σε καμία περίπτωση δεν έρονται και σε, δεν επηρεάζει αυτό τους φόρους που πληρώνουμε σε ευρωπαϊκές χώρες. Επηρεάζει μόνο, αποκλειστικά και μόνο τους φόρους που θα πληρώναμε στη ΗΠΑ. Ε, πρόεδρος, ε, συγγνώμη για το Double Irish και Double Dutch, ε, αυτό το διπλό σύστημα, μπορείτε να το σχολιάσετε. Απάντηση, ναι, να πω για τις Βερμούδες αυτό το ε, σύστημα, αυτή η οντότητα δεν επηρεάζει τα ρόγγελ στα πνευματικά δικαιώματα, διότι έχουμε συμφωνία που συνδυάζεται με το κόστος επιμερισμού που γίνεται μέσα από μια holding εταιρεία ε, στην Ιρλανδία που ε, είναι, το ιδιοκτησιακό καθεστώς είναι Google Inc. Ε, ο κύριος Κόφεντ, ένα λεπτό, διότι πρόσφατα με το Ηνωμένο Βασίλειο συνάψατε συμφωνία για την... μια φορολογική συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο και αν δείτε τα ποσά Μιλάμε για 200 εκατομμύρια λίρες, αν κατάλαβα καλά, από 24 δις, αυτά είναι τα έσοδά σας. Για ε, μια συγκεκριμένη ε, χρονική περίοδο συμφωνήσετε να πληρώσετε αυτά. Δηλαδή αν 0,83 είναι ο συντελεστής, αν κατάλαβα καλά, αν υπολόγισα καλά, για αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο πρώτα απ' όλα θεωρείτε ότι είναι δίκαιο να πληρώνετε στο Ηνωμένο Βασίλειο πρώτον και δεύτερον γιατί ε, συμφωνήσατε για την καταβολή αυτών των φόρων στο Ηνωμένο Βασίλειο ενώ ισχυρίζεστε ότι την τελευταία δεκαετία αυτά που ήδη είχατε κάνει έχουν φορολογηθεί καθόλου για τυπικά εντάξει και βάσει των κείμενων διατάξεων. Γιατί λοιπόν ε, το κάνετε αυτό και το δέχεστε. Ευχαριστώ για την ε, ερώτηση. Ένα λεπτάκι γιατί χάθηκα με το δεύτερο τμήμα, με ζαλίσατε με τη δεύτερη ερώτηση, αν μπορείτε να επαναλάβετε την πρώτη μόνο. Ναι, ρώτησα για το 2010-2015 είχατε 200 δις έσοδα στο Ηνωμένο Βασίλειο και ε, συμφωνήσατε να πληρώσετε 200 εκατομμύρια λίρες σε φόρο. Εάν το υπολογίσετε τελικά καταλήγουμε σε ένα συντελεστή φορολογικό 0,83% για μια συγκεκριμένη ε, περίοδο. Τι να πω, είναι φημισμό το να το χαμηλ, χαρακτηρίσω χαμηλό το συντελεστή. Αυτό ρώτησα. Τι, πιστεύετε ότι είναι δίκαιο. Α, τώρα κατάλαβα, ναι, ναι. Απάντηση. Ε, για τα κέρδη πληρώνουμε και όχι για τα έσοδα πρώτον. Είτε μεγάλη είναι η εταιρεία είτε μικρή. Το κέρδος που μπορεί να αποδοθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο βασίζεται στον αριθμό των εργαζομένων στο Ηνωμένο Βασίλειο, τι επενδύσει που έχουμε κάνει στη χώρα και αυτό πλήρω υπολογίζεται και καταλογίζεται στους λογαριασμού μα. Οι φορολογικέ αρχέ μπορούν να ελέγξουν ε, τους ε, λογαριασμούς ε, που κατατίθενται σε αιτήσια βάση και οι φορολογικές αρχές όπως η HMRC στο Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν και αναδρομικά να ε, ελέγξουν και να διαπιστώσουν αν αυτοί οι λογαριασμοί με το transfer pricing, τη διατιμολόγηση μεταβίβασης για δικαιοδοσίες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο υπολογίζεται με, τη σωστή, με το σωστό τρόπο. Το, αυτό έγινε για έξι χρόνια, εξέτασαν διάφορους παραμέτρους στο Ηνωμένο Βασίλειο, μπορεί να σας φαίνεται μεγαλύτερο. Ξέρετε, είναι αρκετά μακρά η περίοδος και ε, δεν καλύπτουν όλοι οι οικονομικοί έλεγχοι δεκαετία ολόκληρη. Τέλος μου, κατέληξαν στο συμπέρασμα και αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό για ελεγχόμενες πολυεθνικές, ε, είναι ότι ε, τα benchmarks, ε, τα μέτρα που χρησιμοποίησαμε για να υπολογίσουμε επί των κερδών και ο, το, το υπολογισμός του κέρδους αυτή τη συγκεκριμένη δικαιοδοσία ε, δεν, ε, πάντων, για να μην σα τα μπερδεύω, δεν πληρώνουμε επί των εσόδων αλλά επί των κερδών. Ευχαριστούμε. Λέω Πρόεδρος ε, Λούντεκ από το ΕΛΚ για τις δύο ή... Α, μία και για τους δύο ερώτηση. Δύο slots θέλεις δηλαδή. First, one minute. Yeah. One minute. So... Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θα ήθελα ε, να σας πω ποια είναι η άποψή μου για το θέμα. Θεωρώ ότι η κυβέρνηση έκανε λάθος δημιουργώντας ε, ε, ιδιαίτερα περίπλοκες διαδικασίες και νομοθετη... νόμους φορολογικούς, ιδιαίτερα μπερδεμένους και δυνάμια σύνεκτους. Ναι, και ξέρω ότι πολλοί, πολλές εταιρείες χρησιμοποιούν αυτήν την δυνατότητα που δίνεται ε, από ορισμένε ε, κυβερνήσεις ε, έτσι ώστε να προχωρήσουν σε μια ιδιαίτερη, ιδιαίτερα επιθετική φορολογική πολιτική. Προχωράω τώρα στις ερωτήσεις. Πρώτα απ' όλα έχουμε συγκεκριμένε προτάσεις όπως ζήτησε άλλωστε και η εκπρόσωπος της Apple. Ερώτηση ερώτηση λοιπόν. Πιστεύετε ότι τα προγράμματα ε, ε, όσον ε, αφορά την οδηγία η οποία προβλέπει έλεγχο αναχώρα κλπ. Εάν είσαστε έτοιμοι να, και διατεθειμένοι να την εφαρμόσετε. Και επίσης σε σχέση και με την Google να ρωτήσω πώς σκοπεύει να αντιμετωπίσει το θέμα της μόνιμης εγκατάστασης. Ναι, ένα δεύτερο ερώτημα ε, που σχετίζεται με την ανταγωνιστική θέση της, Ευρωπαϊκής, ε, της Ευρώπης. Συγγνώμη. Ε, η άποψή σας είναι μήπως ότι μπορεί να υπάρξουν κάποιες, κάποιες επιπτώσεις αντιθέτου αποτελέσματος. Θα ήθελα να είσαστε σταφίσες στις απαντήσεις σας. Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προτάσεις ε, CCTB της κοινή βάσης δηλαδή θα ε, συζητηθούν συντόμως, θεωρείτε ότι η CCTB μπορεί να αποτελέσει ε, κάποιον, κάποια οδό μείωσης της συμβατότητας και της συμμόρφωσης της φορολογικής ή θα διευκολύνει ακόμα περισσότερο τις εταιρείες σας να προχωρήσουν στις επενδύσεις τους και στις επιχειρήσεις παρατηρήσεις του. απαντήσεις παρακαλώ. Πρώτη ερώτηση, ο εκπρόσωπος της Google. Ε, εμείς ε, είδαμε τις ε, προτάσεις αυτές και φαίνεται ότι πράγματι αντικατοπτρίζουν τις προτάσεις οι οποίες έχουν ξεκινήσει σε διάφορα διεθνή φόρα, κυρίως όσον αφορά την αναχώρα αναφορά. Είναι γεγονός ότι στα τέλη του χρόνου πολλές δικαιοδοσίες φορολογικές θα αρχίσουν να εφαρμόζουν την αρχή αυτή, αλλά βεβαίως θα αποτελέσει μέρος του συνόλου των πολιτικών. Όσον αφορά αφορά τώρα το ζήτημα αυτό που με ρωτήσατε για την μόνιμη εγκατάσταση, εμείς δεν έχουμε ε, κάποια ιδιαίτερη αναφορά όσον αφορά αυτό το θέμα. Δεν μας αφορά στην ουσία και δεν επηρεάζει την ουσία της, ε, της ε, επιχείρησής μας. Ε, εμείς ε, πληρώνουμε ε, φόρους που είναι ίδιοι εάν υπάρχει μόνιμη εγκατάσταση ή όχι. Κοιτάξτε, σε περίπτωση μόνιμης εγκατάστασης ο υπολογισμός των φόρων γίνεται με περίπου τον ίδιο τρόπο που, γίνεται και με το transfer pricing. Δεν έχει κάποια ιδιαίτερη διαφορά. Επίσης, όσον αφορά τώρα την μείωση του κόστους της φορολογικής συμμόρφωσης, αυτό που με ρωτήσατε δηλαδή, πιστεύουμε ότι ναι, οποιαδήποτε διαφοροποίηση ε, καθεστώτων μεγάλη θα δημιουργήσει όντως μεγαλύτερο ε, πρόβλημα ως και μεγαλύτερο κόστος όσον αφορά αυτή τη συμμόρφωση, πράγμα βεβαίως οξύμορο, εάν λάβει κανείς υπόψη ότι συζητούμε πάντα για ελευθερία κυκλοφορίας, ελευθερία διακίνησης, ελευθερία μόνιμης εγκατάστασης οπουδήποτε. Όσον αφορά το, το επανειλημμένα ε, την κοινή βάση, ε, επανειλημμένα ε, έχει συζητηθεί το θέμα αυτό και νομίζω ότι όσο πιο σαφείς είναι οι κανόνες τόσο καλύτερα για όλους. Απάντηση από πλευράς της Apple. Όσον αφορά την ε, ε, διεθνή φορολογική μεταρρύθμιση πρέπει να σας πω ότι εμείς έχουμε ξεκινήσει ήδη ε, να προετοιμαζόμαστε κυρίως όσον αφορά την πολυμερή προσέγγιση οι αρχές είναι πολύ σημαντικό να είναι ίδιες και αυτό είναι εξίσου σημαντικό με την απλούστευση. Θα πρέπει να είναι απλή η νομοθεσία. Όσον αφορά τις, ε, την, ε, τα μέτρα τα οποία προτείνει η ε, οδηγία για την φορολογική αποφυγή, ναι, θεωρούμε ότι τα όσα περιέχονται σε αυτήν την ε, οδηγία, κυρίως όσον αφορά τη σαφήνεια του BEPS, ε, είναι ε, πολύ σημαντικό. Απλώς, πολύ, βεβαίως, πολύ σημαντική είναι και η σωστή υλοποίηση και εφαρμογή των αρχών αυτών η σαφήνεια ε, και η απλότητα θα βοηθήσει την σωστή εφαρμογή ε, των φορολογικών ρυθμίσεων ε, και καθεστώτων αλλά βεβαίως θα πρέπει να υπάρξει και ισοτιμία όλων όσον αφορά την CCTB, CCCTB ε, ναι είναι γεγονός ότι ε, μπορεί να απλουστεύσει την φορολογική βάση και αν αυτό γίνει όντως θα είναι ε, πιο θετικά τα πράγματα. Αλλά για την ώρα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. I guess the simpler the better. Simpler the better. <laughs> okay. Uh, on behalf of... Από τους σοσιαστές και δημοκράτες, ο Πέτερ Ζήμων. Τι στόχο έχετε εσείς και, και τους δύο. <laughs> Ποιον έχετε στο στόχαστρο, ναι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η πρώτη ερώτηση είναι στη Google. Με διέφερα αυτό που άκουσα ότι τηρείτε τους κανόνες. Πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε. Με τις ε, Βρετανικές φορολογικές αρχές συμφωνείτε να πληρώσετε 172 εκατομμύρια από τους χρωστάτε και περίπου τα ίδια στην Ιταλία και στη Γαλλία. Στην Ιταλία διαβάζουμε για κάτι για 200 εκατομμύρια ευρώ συνολικά. Εγώ τώρα τι να συμπεράνω, ότι στο παρελθόν δεν ήταν τόσο άψογη η φορολογική σας συμπεριφορά. Ε, είναι εργατικό ατύχημα. Δεύτερη ερώτηση. Η δοντολογία της επιχείρησης. Κοιτάω τις 10 αρχές που διέπουν την εταιρεία. Είναι τέλεια αυτά. Στο 6 λέτε να κερδίζουμε χρήματα χωρίς να ζημιώνουμε κανέναν. Έτσι όπως τα λέτε είναι απόλυτο θεμητά να εκμεταλλεύεστε τους φορολογικούς κανόνες και να πληρώνετε φόρους που είναι ένα κλάσμα εκείνων που κανονικά πληρώνουν οι εθνικές εταιρείες. Αυτό ανταποκρίνεται ε, στον κανόνα σα, στο δεκάλογο των αριθμών 6, να βγάζετε λεφτά χωρί να ζημιώνετε κανέναν. Δεν ζημιώνεται το γενικό σύνολο μαζικά. Και το βλέπουν αυτή τη στιγμή και το ακούνε live σε όλη την Ευρώπη από το web stream οι πολίτες και παρακαλώ να τους εξηγήσετε. Ευχαριστώ. Ο Κοέν. Ευχαριστώ. Όπως σας είπα προηγουμένω, είναι κοινή πρακτική για τις φορολογικές αρχές να ζητούν από τις εταιρείες να ελέγξουν τους λογαριασμούς τους ε, ε, αναδρομικά για να δουν ε, τι μέθοδο είχαν και πώς έκαναν τις μεταβιβάσεις. Ποιες ήταν οι μέθοδοι και τα benchmark που χρησιμοποιούσαν για να και τα κέρδη σε κάποια δικαιοδοτική περιφέρεια. Τι συμπεριλαμβάνεται, τι εξαιρείται. Στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι μια διαδικασία που καλύπτει ένα μακρύ χρονικό διάστημα, μακρύτερο από ό,τι αλλού. Σας το είπα και προηγουμένως. Και νομίζω ότι ο στόχος είναι ότι το Ρέμι Βασιλείο ήταν από τις πρώτες ε, ε, χώρες ε, που κοίταξαν πώς είναι διαφορετική η κατάσταση της ψηφιακής οικονομίας και της εταιρεία τους σε σχέση με τις υπόλοιπες εταιρείε. Έγινε μια προσαρμογή προς τις φορολογικές μας υποχρεώσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό είναι πάρα πολύ φυσιολογικό για μια πολυεθνική. Για άλλες χώρες είδα ε, κάποια δημοσιεύματα και εικασίες, αλλά στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι το μόνο που έχει λήξει. Για τη διοντολογία είναι σημαντική ερώτηση και μπαίνει όταν συζητούμε για νομοθετικές αλλαγές και ποιο είναι το νομικό πλαίσιο που θέλουμε να έχουμε για τη φορολογική πολιτική. Πώς θα πρέπει να λειτουργεί ένα φορολογικό σύστημα. Αυτό είναι θέμα και ηθικό και δεντολογικό. Αυτή τη στιγμή ε, οριστούν οι κανόνες, οφείλουν οι εταιρείε να τους στηρούν. Και όταν πληρώνουμε ένα πυροελάχιστο κλάσμα ε, σε σχέση με τι πληρώνουν άλλε εταιρείε, αυτό δεν ευσταθεί καθόλου. Αν δείτε συνολικά, 19% πληρώνουμε τα τελευταία χρόνια και 20% ε, ε, πληρώνουν και άλλες πολυεθνικές. Ναι, δεν ρώτησα αυτό όμως, συμπληρωματική προς τον συνάδελφο από την Google. Ναι, ακούστε με. Είναι ηθικό και δεντολογικό να συγκρίνεστε με άλλους και να λέτε ότι είμαι στο ίδιο φάσμα οπότε εντάξει είμαι. Εσείς ε, δεσμεύεστε ε, και έχετε ένα δεκάλογο ε, για ηθική και δεντολογία στην επιχείρησή σας και είναι εντάξει να πληρώνετε ένα κλάσμα των φόρων που πληρώνουν άλλες εταιρείες μικρομεσαίες, εθνικό επίπεδο, όχι πολυεθνικές. Το θεωρείτε σωστό να συμμετέχετε μόνο κατά ένα κλάσμα στο γενικό ε, κοινό καλό, ε, πολύ λιγότερο από κάθε ε, κανονικός φορολογούμενος. Εμείς πληρώνουμε όπως όλες οι άλλες εταιρείε στις χώρες που δραστηριοποιούμαστε. Και αν συγκρινόμαστε με άλλες εταιρείε, όχι. Θέλω να το διορθώσω. Δεν είναι καθόλου κλάσμα αυτό που πληρώνουμε. συγκρινόμενοι με άλλες εταιρείε. Δεν ισχύει αυτό. Ένα από τα πράγματα που μπορούμε σήμερα, ελπίζω να κάνουμε, είναι να συζητήσουμε επί της ουσίας, με γεγονότα και πραγματικά περιστατικά. Είναι πολύ σημαντική η συζήτηση αυτή που γίνεται εδώ για το πώς τηρούμε τους κανόνες. Εταιρείε και μεταξύ αυτών η Google ε, επιζητούν την ε, συμμόρφωσή τους, θέλουν να είναι νομοταγείς. Αλλά ε, τους κανόνες δεν τους γράφουμε εμείς. It's whether it's fair or unfair. that's clear. Μάλιστα, ε, να ε, προσέχουμε και το χρόνο. Μπέρντ Λούκε, εξ ονόματος των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών. Η ερώτησή μου απευθύνεται στην εκπρόσωπό της Apple. Ερώτηση πρώτη. Ένας εκπρόσωπος της εταιρείας σας πήγε στην υποβιτροπή της Γερουσίας των ΗΠΑ και είπε ότι οι ειδικέ φορολογικές κατασκευές στην Ευρώπη το Double Irish και το Dutch Sandwich μάλλον ε, ε, εννοούσε στα Βρετανικά παρθένα νησιά ε, χρησιμοποιείται για να κάνει έρευνα η εταιρεία στις Ηνωμένε Πολιτείε και να τη χρηματοδοτήσει εκεί. Αυτό είναι κρατική ενίσχυση ή τίποτα άλλο. Apple. Γιατί η Ευρώπη χρηματοδοτεί δηλαδή έτσι ε, την ερευνητική δραστηριότητα και την καινοτομία στις ΗΠΑ της Apple. Και μια σύντομη ε, ερώτηση να απαντήσω σε αυτό που απαντήσατε εσείς. Αυτή η φορολογική κατασκευή που σας ανέφερα στην Ευρώπη έχει ε, επιτρέψει μία νόμιμη φοροαποφυγή και το τονίζω νόμιμη φοροαποφυγή στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Η κυρία Θα ήθελα να απαντήσω στο πρώτο κομμάτι και μετά η Τζούλη στο τελευταίο Μιλήσατε για τις ακροάσεις στη Γερουσία, τον είπα. Πρώτα απ' όλα, δεν έχουμε διπλή δομή Irish ε, ε, έχουμε συνέπεια στην ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουμε και γι' αυτό ε, καθοδηγούμαστε κεντρικά, κυρίως από τη ΣΥΠΑ. 70.000 ε, εργαζόμενοι στη ΣΥΠΑ, τους περισσότερους φόρους εκεί τους πληρώνουμε. πληρώνουμε βεβαίως και για τα τοπικά υποκαταστήματα βάσει της φορολογικής νομοθεσίας στις χώρες. Δεν έχουμε μία διπλή τέτοια Ιρλανδική δομή. Από όσο ξέρω ε, ε, διακόπτει ο κύριος Λούκο. Δεν θέλω να συζητήσουμε στις λεπτομέρειες τι σημαίνει Double Θέλω να σχολιάσετε αυτά που είπε ο εκπρόσωπός σα στη Γερουσία. Ότι οι φορολογικές ρυθμίσει ε, στην Ευρώπη χρηματοδοτούν την έρευνα και ανάπτυξη της Google στη ΣΥΠΑ. Η φορολογική απάντηση. Ε, οι φορολογικές ρυθμίσεις στην Ευρώπη χρηματοδοτούν την έρευνα και ανάπτυξη. Αυτό μου λέτε ότι είπε. Εγώ αυτό θυμάμαι, λέει ο κ. Λουκ. Λοιπόν, ε, θα ήθελα να πω, δεν είναι, έχω γνώση τέτοιες δήλωσες, ε, πληρώνουμε του, του, τα, τους φόρους μας στη ΣΥΠΑ, δηλαδή υπάρχει μεταφορά των φορολογικών υποχρεώσεων στη ΣΥΠΑ, αυτό ναι και χρειαζόμαστε για τα νέα εργαλεία, για την έρευνά μας, για την ανάπτυξη νέων εργαλείων, για τα νέα καταστήματα και ούτω καθεξής. Δεν πιστεύω λοιπόν ότι αυτό εννοούσε, ότι έγινε τέτοια δήλωση από εκπρόσωπό μας. Το τελευταίο που είπατε, Τζούλια, σας παρακαλώ να ε, επεκταθείς για αυτά τα περί φορολογικών δομών. Λοιπόν, ε, πώς ε, λειτουργούμε στην Ιρλανδία. Ανέκαθεν ήταν μια εταιρεία που δεν έχει εκεί φορολογική έδρα. Νομίζω ε, σε αυτό ε, να αναφερόσασταν ότι μέσω ε, cost sharing ε, τελικά χρηματοδοτούμε την έρευνα στη ΣΥΠΑ. Εγώ, ε, λέει ο κύριος Λουκ, με οποιαδήποτε δομή και να έχετε στην Ευρώπη, Όμω αποφεύγετε τους φόρους εδώ και χρηματοδοτείτε την έρευνα στη ΣΥΠΑ. Απάντηση. Δεν έχουμε καμία τέτοια δομή στην Ιρλανδία αλλά και σε υπόλοιπε ευρωπαϊκές χώρες όπου πληρώνουμε φόρους αναλογικούς με τη δραστηριότητα που διεξάγονται σε εκείνες τις χώρες, τίποτα παραπάνω. Λουκ, μπορείτε να μου εξηγήσετε γιατί θεωρείτε ότι δεν έχετε αποφύγει ε, τη φορολόγηση ενώ ο συντελεστής είναι 12,5 στην Ιρλανδία και εσείς πληρώνετε 2%. Δεν είναι φοροαποφυγή. Μα απάντηση, εμείς πληρώνουμε τον συντελεστή που προβλέπετε 12,5 στην Ιρλανδία αλλά δεν έχουν φορολογική έδρα οι, οι, οι θηγατρικές μας ε, στην Ιρλανδία και άρα πληρώνουμε επί των κερδών ε, στην Ιρλανδία μόνο για τις δραστηριότητες ε, που διεξήχθησαν στην Ιρλανδία και βάσει του αριθμού των υπαλλήλων και γραφείων που έχουμε εκεί. αυτά υπάγονται μόνο στην Ιρλανδική φορολογία και φυσικά πληρώσαμε πλήρως το συντελεστή 12,5%. Ευχαριστούμε. Ραμόν Τρεμόσα, Άλντε. Ευχαριστώ. Ραμόν. σε ποιον, σε ποιον υπόβαλε το ερώτημα. Άντα μου κάνει καλώ ορίσατε στο Κοινοβούλιο. Ε, χαίρομαι που σα ξαναβλέπω. Πριν από ένα χρόνο μιλάγαμε για την, το, την αντιτράστ ε, επιχείρηση της ε, που σχετιζόταν με την Google. Ελπίζουμε να δεχτείτε τις προσκλήσεις που θα σας στείλουμε και φέτος, γιατί τρία χρόνια σας κυνηγάμε να έρθετε, ε, χαιρόμαστε που επιτέλους ήρθατε. Ε, θα ήθελα για τα φορολογικά ζητήματα για την Google μια σύντομη ερώτηση να σας κάνω. Πρώτον, διάβασα στον τύπο ότι σχεδόν 12 δις κέρδη ε, τα στείλατε της Βερμούδες από τη πλευρά ε, Google. Ε, αληθεύει. Δεύτερον, ε, κάνατε συμφωνία με την Αμερικανική κυβέρνηση και μετά και με τη Γαλλική για να πληρώσετε κάποιους φόρους σε αυτές τις χώρες. Η επόμενη ποια θα, κυβέρνηση θα είναι της Ιταλίας. Μπορείτε να μας ενημερώσετε. Και τέλος. Ε, η Google στην Ευρώπη περνάει το μήνυμα ότι βοηθάει τις μικρομεσαίες. Ε, πολύ μου αρέσει το σύνθημά σας, αλλά έχω την εντύπωση ότι υπερφορολογούνται οι μικρομεσαίες στην Ευρώπη διότι οι πολυεθνικές δεν πληρώνουν τους φόρους τους στην Ευρώπη. Άρα το μέρος του φορολογικού βάρους που τους αναλογεί είναι δυσανάλογα μεγάλο. Βαραίνει κυρίως τις μικρομεσαίες. Μηπω, θα μπορούσατε κι εσείς να επιμεριστείτε, να υπομειστείτε συγγνώμη, ένα μέρος αυτής της ευθύνη για να υποστηρίξετε και τις κοινωνικές υπηρεσίες παρέχοντα στην Ευρώπη. Και το θέμα δεν είναι αν είναι σύνομο ή έκνομο αυτό που κάνετε. Το ζήτημα είναι αν ε, είναι fair, αν είναι ισότιμη όρια ανταγωνισμού. Ε, και εγώ χαίρομαι που σας ξαναβλέπω. Όσον αφορά αυτά τα 12 δις, δεν είμαι απόλυτα ε, σίγουρος τι διαβάσατε ως δελτίο τύπου, αλλά πρέπει να σας πω ότι τα χρήματα τα οποία καταλήγουν ε, στις ε, Βερμούδες είναι χρήματα τα οποία έχουν ήδη φορολογηθεί ε, στην Ευρώπη και Όσον αφορά το Ηνωμένο Βασίλειο και αυτό που είπατε για άλλες χώρες, η μόνη δικαιοδοσία με την οποία έχουμε κάνει ε, κάποια συμφωνία είναι το Ηνωμένο Βασίλειο και μόλις ολοκληρώθηκε η συμφωνία ε, την κοινοποιήσαμε και την δημοσιοποιήσαμε. Ε, εάν υπάρξουν παρόμοιες ρυθμίσεις σε άλλες δικαιοδοσίες ε, θα τις δημοσιεύσουμε επίσης. Όσον αφορά το θέμα με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, χαίρομαι που το θίξατε γιατί όντως εμείς, έχουμε, εμείς λειτουργούμε βάσει ενός σχήματος που εμπλέκει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις γιατί θεωρούμε ότι είναι ο καλύτερος τρόπος για να φτάσουμε στους καταναλωτές σε ολόκληρο τον κόσμο με τον τρόπο αυτό έχουμε επιλέξει γεωγραφικά και λοιπά να προσεγγίζουμε τους ε, πελάτες. Τώρα όσον αφορά τον σωστό επιμερισμό, δίκαιο επιμερισμό του φορολογικού άχθους ε, Κοιτάξτε, από τη στιγμή που ε, η μία εταιρεία είναι κερδοφόρα, τότε οπωσδήποτε πληρώνει ε, φόρους. Ε, και ξέρω ότι όταν κάποια εταιρεία είναι μικρομεσαία και έχει ε, ένα συγκεκριμένο ποσοστό κερδοφορίας, τότε έχει και έναν ειδικό φορολογικό συντελεστή. Πρέπει να σας πω ότι εμείς πληρώσαμε την προηγούμενη χρονιά 56 εκατομμύρια δολάρια και θεωρώ ότι είναι σημαντικό. Ναι, ενδεχομένως και άλλες ε, χώρες, λέει ο Πρόεδρος, θα βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις ε, με την Google, μεταξύ των οποίων ε, και η Γαλλία, γιατί οι εκεί εκπρόσωποι τη εταιρεία ζητούν διαδικασία αντίστοιχη με αυτή της, του, μεγάλου, του Ηνωμένου Βασιλείου. Φάβιο Μάζη. Αρχίσω από το ίντερνετ και μετά θα πάω στο iPhone. Δηλαδή, Google πρώτα έχετε holdings στις κάτω χώρες που πληρώνετε πολλά λόγια από την Ιλανδία αυτό το sandwich που λέγαμε και σύμφωνα με την ενημέρωσή μου ε, στις κάτω χώρες ε, ε, απασχολείται ακριβώς μηδέν ε, υπαλλήλους. Δηλαδή με ένα τηλεφωνητή πόσα κέρδη βγάζετε και πόσα, ποια είναι η οικονομική δραστηριότητα. Από το 2009 η Google ε, έχει αναφέρει 25 ε, ε, θηγατρικές ε, στις ΗΠΑ και έκτοτε έχουν μειωθεί στις δύο στην Ιρλανδία. Πού είναι οι 23 που λείπουν οι θηγατρικές. Το Μάρτιο του 2012 ήταν ακόμα ενεργές. Μπορείτε να μας πείτε τι έχουν γίνει αυτές οι 23 από το 2009 μέχρι σήμερα και που βρίσκονται σε ποιους παραδείσους και πώς λειτουργούν. Και γιατί έχετε επιλέξει να μην τα δημοσιεύετε πλέον αυτά. Uh, σε ό,τι αφορά το Google Netherlands, είναι ένα holding πραγματικά. Ε, ε, ανήκει σε αυτή τη ε, ρύθμιση της Βερμούδας που δεν έχει να κάνει με τα όσα οφείλουμε ως φόρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά στις Ηνωμένε Πολιτείες. Σε ό,τι αφορά την ουσία στις κάτω χώρες έχουμε μια μετρική εταιρεία που έχει 200 εργαζομένους, κάνει και όλες τις δουλειές μας και πληρώνει και φόρους. Και τις επενδύσεις και τους υπαλλήλους ε, το υπολογίζουμε και είναι ουσιαστικά... Ναι, αλλά έχετε μηδέν υπαλλήλους ως Google. Ναι, ε, σας είπα ότι είναι ε, μια εταιρεία που πληρώνει φόρους. Θέλω να επισκεφθώ πάρα πολύ τα γραφεία σας. Θα ήταν συναρπαστικό. Με χαρά να έρθετε και στην Ελλάδα και στις κατοχώρες και όπου θέλετε. Όπως σας είπα, το φορολογικό σύστημα των πολιτείων είναι διαφορετικό από τα άλλα. Ε, έχει την επικράτεια που επιβάλλει ε, το φόρο. Μπορεί να σας φαίνεται περίπλοκο ή περίεργο, αλλά σύμφωνα με το Διεθνή Φορολογικό Κώδικα, το σύστημα αυτό δεν έχει να κάνει με το τι ε, πληρώνουμε στην Ευρώπη, αλλά τους φόρους που οφείλουμε στις Ηνωμένες Και αυτή τη μελέτη που είπατε για τις θηγατρικές ε, σε φορολογικούς παραδείσους. Δεν την έχω δει αυτή τη μελέτη, με χαρά να τη δω και να την ε, διαβάσω κι εγώ. Είναι πάρα πολύ δημόσια τα στοιχεία που δραστηριοποιούμαστε και το θέμα των Βερμούδων έχουμε την έδρα μας στην Ιρλανδία, όλα αυτά είναι δημόσια, δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε και δεν νομίζω να αλλάζει τίποτα, ούτε να έχει αλλάξει ουσιαστικά από το 2009. Και πώς έχει και παραέχει και είμαι βέβαιος ότι θα ξανάρθει, θα μας τα ξαναπείτε αυτά. Ε, η ερώτηση στην Apple. Ο συνάδελφος από την Google μόλις μίλησε για το αμερικανικό φορολογικό σύστημα, όπου πληρώνεις μόνο φόρους αν έχεις επαναπατρίσει κέρδη 200 δις ε, δολάρια έχει πληρώσει εκτός της, ε, των Ηνωμένων Πολίτων και μιλήσατε για ελαφρύνσεις ε, στο Αμερικανικό σύστημα τι πληρώσατε το 2014 και 2015 ως φόρο επιχειρήσεων γιατί με την η Ιρλανδική σας δομή εκεί δεν ε, έχουμε ε, σαφή στοιχεία από τους λογαριασμούς. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέτε επιλεκτικά συζητάει με αμερικανικές ε, πολυεθνικές. Δηλαδή νομίζετε ότι δεν έχει άλλη δουλειά να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σπαταλάει εκεί το ανθρώπινο δυναμικό της να ασχολείται με τέτοια πράγματα. Παρακαλώ, κυρίες. Um, Πρώτη ερώτηση που σχετίζεται με το αμερικανικό φορολογικό σύστημα και τη φορολογική μεταρρύθμιση. Ζητούσαμε τη φορολογική μεταρρύθμιση και έχουμε κάνει και σχετικές δηλώσεις. Θέλουμε ε, μείωση του εταιρικού φόρου στη ΣΥΠΑ γιατί είναι και από τους υψηλότερους συντελεστές ε, στον κόσμο. Θέλετε δηλαδή να πάρετε πίσω και λεφτά μετά τη μεταρρύθμιση. Θεωρούμε ότι είναι σκοπιμότερο και ευνοϊκότερο για μας να είναι χαμηλότερος ο συντελεστής ε, μετά τη μεταρρύθμιση. Μας ρωτήσατε πόσο φόρο έχουμε πληρώσει. Όπως είπε η Κάση, νομίζω ότι είμαστε από αυτούς που πληρώνουν τα περισσότερα στον κόσμο από το 2015. 13,2 δις σε φόρους παγκοσμίω πληρώσαμε. 26,4 ήταν ο μέσο όρος του φορολογικού συντελεστή που πληρώσαμε. Μιλήσατε, ε, μας ρωτήσατε για του φόρου που πληρώσαμε στην Ιρλανδία. Δημοσίω δεν το κοινοποιούμε. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση σα ρώτησα, όχι για τι 28 χώρε, όχι μόνο για την Ιρλανδία. Δεν ε, κοινοποιούμε αυτό, δεν έχουμε υποχρεώσεις ε, κοινοποίησης για τους φόρους που πληρώνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οπότε δεν είναι δημόσια διαθέσιμη αυτή η πληροφορία, θεωρείται εμπιστευτική. Ε, προστατεύεται. Είναι δικαίωμα του φορολογουμένου, αν θέλετε, να μην κοινοποιεί τις πληροφορίες αυτές. Εκτός ε, μικροφώνου σχόλια. για την υποβολή εκθέσεων ε, αναχώρα στα πλαίσια του BEPS μπορεί να αλλάξει αυτό. Όταν θα αρχίσουν να ισχύουν αυτές, αυτοί οι κανονισμοί θα υποβάλουμε και εμείς τα στοιχεία μας. Σε χώρες ε, που έχουμε δημόσιες πληροφορίες, τις έχουμε. Συγγνώμη, αλλά δεν απαντήσατε στην τελευταία μου ερώτηση. Εγώ ζητώ συγγνώμη, λέει πρόεδρος. Ε, ε, κύριε Ντεμάζη, δεν έχετε άλλο χρόνο. Μόλις κάτω από τη Ευχαριστώ. Το σύνθημα της Google... Για την Google. Μόνο στην Google απευθύνεστε. Ναι. Ε, μην είστε κακοί. Αυτό είναι το σύνθημα της ε, Google και το αλλάξανε τώρα, πρέπει να το αλλάξουμε, κάντε το σωστό. Ε, θα πρέπει λοιπόν να ντρέπεστε από την ε, κατακραυγή με τη συμφωνία που κάνετε με την HMRC, η φορολογική αρχή στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τζον Μακδόναλ, ε, ο Υπουργό Οικονομικών, είπε στο Financial Times ότι έγιναν και κλειπέων το θηρόνι οι διαπραγματεύσει και δεν αρμόζει να εφαρμοστεί τέτοια συμφωνία γιατί είναι δυσανάλογο για του υπόλοιπου φορολογουμένου. Αυτό νομίζω είναι επιζήμιο όχι μόνο για το, την παρουσία σα στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και στην Ευρώπη. Ε, λέτε ότι συμμορφώνεστε με το νομοθεσία και καταβάλλεται τους φόρους ε, όπως ε, ε, προβλέπετε. Ε, αυτό ισχυρίζεται και σήμερα και λέτε ότι θέλετε μεταρρύθμιση φορολογική τη ΕΠΑ και αυτό θα ήταν καλό για εσά γιατί πλήττεται η φήμη σα ακόμη και με αυτέ τι ε, σύνομε δραστηριότητε με τι οποίε όμω όντω φοροδιαφεύγεται. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω εσά, Google, νομίζω ισχύουν και για τι δύο εταιρείε, οι εταιρείε. Λοιπόν, να σα ρωτήσω το εξή. Ξαναλέω με το σύνθημα κάνε το σωστό. Ε, ε, τι πιστεύετε λοιπόν για την πλήρη κοινοποίηση στοιχείων αναχώρα country by country reporting. Στη συνέχεια, ε, για την κοινή ενοποιημένη βάση. Κάποια κράτη-μέλη μπλοκάνουν τη διαδικασία, όπως μάλλον θα ξέρετε, στο Συμβούλιο. Και από ό,τι φαίνεται ότι είναι καλύτερες οι διαπραγματευτικές ικανότητες για αυτές τις συγκεκριμένες κυβερνήσεις. Μπορείτε να προχωρήσετε, παρακαλούμε, το θέμα της CTB στο Συμβούλιο. Ευχαριστώ, Διευθυντής. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας όσον αφορά τα διοντολογικά ζητήματα κλπ. Κοιτάξτε, πιστεύω ότι αυτό είναι θέμα που πρέπει να εντάσσεται στην συμμόρφωση ε, και πιστεύω ότι είναι θέμα φορολογικής πολιτικής και θα πρέπει να ε, ληφθεί υπόψη κατά αυτή την έννοια. Η ε, συμμόρφωση προς, τους φορολογικούς, προς τις φορολογικές νομοθεσίες είναι απολύτως απαραίτητη. Εμείς και στην Ιρλανδία θέλουμε σαφείς κανόνες με τους οποίους να μπορούμε να συμμορφωνόμαστε ε, δεν μας ενδιαφέρουν και δεν θέλουμε ε, καταχρηστικούς φόρους ε, ή θέλουμε μια λογική φορολογική για να ξέρουμε και εμείς τι πρέπει να εφαρμόσουμε και τι, με τι πρέπει να συμμορφωθούμε. Όσον αφορά τώρα τους δημοσιοποιημένους φόρους, εμείς αναδικαιοδοσία στην οποία λειτουργούμε δημοσιοποιούμε τους, ε, τα φορολογικά μας ε, στοιχεία και τους ε, φόρους που πληρώνουμε. Όσον αφορά το κατά πόσον θα μπορούσαμε να στηρίξουμε την κοινή ενοποιημένη βάση CCCTB, όπως είπα και προηγουμένως, Εάν αυτό δώσει ε, μεγαλύτερη συνεκτικότητα και μεγαλύτερη διαφάνεια στους ε, ε, νόμους, ναι, θα μπορούσαμε, ναι, θεωρούμε ότι θα είναι θετικό στοιχείο. Τώρα, όσον αφορά την HMRC, είναι μια αυστηρά ανεξάρτητη αρχή ε, μας ήλεγξε. Ε, στην διαδικασία υπήρξαν τρεις φάσεις ε, και υπήρξαν πάρα πολλοί και ενδελεχείς έλεγχοι και στο τέλος στάσαμε σε μια συμφωνία η οποία βέβαια προϋπέθεσε και μια, μια μεγάλη προσπάθεια και από τη δική μας πλευρά. Επαναλαμβάνω είναι μια ανεξάρτητη αρχή με την οποία ήρθαμε σε μια συμφωνία να κάνω επιπλέον ερώτηση. Θα ήθελα να μου πείτε την άποψή σας ε, για την διαφάνεια. Δηλαδή λέτε ότι θα εφαρμόσετε το νόμο. Ε, ε, πιστεύετε όμως ότι δεν πιστεύετε ότι θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια όχι μόνο όσον αφορά του πόσους φόρου πληρώνετε αλλά και όσον αφορά τα εισοδήματά σας επί των οποίων πληρώνετε φόρους ε, και σχετικά με το CCCTB έχετε ήδη κάνει κάποια εργασία, έχετε κάνει κάποια πρόταση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχετε κάνει υπολογισμό αν θα πληρώνετε λιγότερα ή περισσότερα σε σχέση και αν εφαρμοστεί αυτό. Απόφαση. Απάντηση. Θεωρώ ότι πληρώνουμε το σωστό ε, ε, ποσοστό φόρου όσον αφορά τώρα την αναχώρα αναφορά. Ε, υπάρχουν ενδεχομένως πληροφορίες οι οποίες έχουν κάποιον ευαίσθητο εμπορικό χαρακτήρα και ίσως δεν θα έπρεπε να δημοσιοποιούνται. Υπάρχουν ας πούμε κάποια κόστη τα οποία αφορούν συγκεκριμένα benchmarks ή συγκεκριμένη έρευνα κτλ. Όντως υπάρχουν κάποιες ε, πληροφορίες οι οποίες ε, καλύπτονται από το φορολογικό απόρριτο ε, και ίσως αυτό είναι καλό. Όσον αφορά τώρα το CCTB. δεν γνωρίζω όλους τους κανόνες τους οποίους θα εισαγάγει αλλά οπωσδήποτε θα είμαστε και υποχρεωμένοι να συμμορφωθούμε γιατί εμείς πάντα ακολουθούμε αυστηρά τις υποχρεώσεις μας. Thank E ο Μάρκο Τζάνι. Θα ήθελα και στους δύο να κάνω ερωτήσεις. Πολύ ωραία. Η πρώτη μου ερώτηση αφορά τον εκπρόσωπο της Google. Θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο για αυτά τα 11 ε, ε, δις ε, ευρώ τα οποία φαίνεται ότι σύμφωνα με δημοσιεύματα μετακινήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς, την Βερμούδα, προς τις Βερμούδες. Φαίνεται ότι υπήρξε κάποια συμφωνία σε σχέση με ενδεχόμενη καταβολή κάποιου τμήματος των φόρων στην Ολλανδία. Από την άλλη πλευρά εσείς μας είπατε ότι είστε παρόντες σε κάποια Κάποιε χώρε στις οποίες έχετε δραστηριότητες με μεγάλη προστιθέμενη αξία και βοηθάτε και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις κτλ. Δεν καταλαβαίνω όμως ποιε είναι αυτές οι δραστηριότητες ε, ε, προστιθέμενης αξίας ε, ποιε είναι αυτές που έχετε στην, στις βερμούδες έτσι ώστε να μετακινήσετε προς τα εκεί 11 δις ευρώ σε σχέση τουλάχιστον με δραστηριότητες που έχει η Google στην Ολλανδία ή στην Ιρλανδία. Αυτή είναι η πρώτη μου ερώτηση. Κύριε Διευθυντά παρακαλώ. Όπως είπα και προηγουμένως και όπως και ο συνάδελφος Νίκος Λάμπερ, ο συνάδελφός μου σας είχε πει το Δεκέμβριο, δεν έχουμε έδρα στην Βερμούδα. Αυτή η δομή ε, στις Βερμούδες είναι ε, ε, σχετική με, μία, με, κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που, έχουν, που έχει η φορολογική δομή στις Ηνωμένε Πολιτείες. Αυτό που ονομάζουμε εμείς κανονική παρουσία είναι εκεί που έχουμε παρουσία και εργαζόμενους. Ε, ε, τώρα η παρουσία μας ε, στις Βερμούδες είναι ένας τρόπος να αντιμετωπίσουμε και να εφαρμόσουμε κάποιους νόμους και κάποιους κανόνες τους οποίους εφαρμόζουν και άλλες εταιρείες παντού και στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη. για να συμπληρώσω αυτά που μόλις υπόθηκαν έτσι ώστε να το κατανοήσουν όλοι οι συνάδελφοι και θα με διορθώσετε εάν σφάλω. Θα πρέπει να κατανοήσουμε το σύστημα ε, των πολυεθνικών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Για τα κέρδη τα οποία έχουν ε, γίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες ε, φορολογούνται επιτόπου. Τώρα, για κέρδη πολυεθνικών σε άλλες χώρες τότε θα πληρωθούν οι φόροι αλλού γιατί το αλλού μπορεί να σημαίνει οτιδήποτε μπορεί να σημαίνει και κάποια φόρο αποφυγή ή κάποια μόχλευση ε, φορολογική. Εμένα δεν με ενδιαφέρει σε αυτή την περίπτωση, το κρίνετε εσείς αν είναι σωστό ή όχι. Σε αυτή την περίπτωση λέω τα χρήματα πηγαίνουν στις Βερμούδες έτσι ώστε να μπουν στη διαδικασία deferral. Δηλαδή δεν θεωρούνται, δεν θεωρείται καθαρό φορολογικό, ε, προηγούμενο συγγνώμη κέρδος. Τουλάχιστον αυτό συμβαίνει σύμφωνα με τις αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών. Έτσι δεν είναι, ναι, ευχαριστώ πρόεδρε, λέει εκπρόσωπος της Google. Ερώτηση για την Apple. Ε, στην εκπρόσωπο της ε, Apple ε, ήθελα να κάνω μια πρώτη ερώτηση η οποία αφορά κάποια στοιχεία ε, σχετικά με το πόσο ξοδεύεται κάθε χρόνο ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολο. Εάν έχετε δηλαδή κάποια στοιχεία όσον αφορά τις, ε, την, τις φορολογικές συμβουλές τις οποίες λαμβάνετε για τις φορολογικές σας δηλώσεις ας πούμε και τη φορολογική συγκατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πόσα πληρώνετε και επίσης πόσα πληρώνετε στην, Ευρωπαϊκή στην πόσα πληρώνετε στις Ηνωμένες Πολιτείες έτσι ώστε ε, να έχετε βελτιστοποίηση των φορολογικών. Ε, ε, στην Ιταλία φαίνεται επίσης ότι έχετε μία διαδικασία ξεκινήσει όσον αφορά μη όσον αφορά κέρδη μη δηλωθέντα. Βεβαίως εσείς μας είπατε ότι αυτά γίνονται μέσα στα πλαίσια του transfer pricing, της τιμής μεταβίβασης, αλλά δεν θεωρείτε ότι ότι εδώ προκύπτει κάποιο δεοντολογικό ζήτημα γιατί ενδεχομένως όλες οι εταιρείε θα μπορούσαν να ε, χρησιμοποιούσουν αυτήν την διαδικασία transfer pricing έτσι ώστε και ευελπιστώντας ότι δεν θα τους τσακώσει κανείς. Παρακαλώ. Ρωτήσατε πόσα δαπανούμε για φοροτεχνικούς και παροχή συμβουλών. Δεν έχω αυτά τα στοιχεία να σας δώσω, τα αριθμητικά ετησίως, αλλά νομίζω και επίσης ότι δεν τα δημοσιοποιούμε. Καλά, γραπτός μπορείτε να απαντήσετε, δεν πειράζει. Ε, χρησιμοποιούμε συμβούλους για διάφορα πράγματα, για όλες τις δραστηριότητες μας σε κάποιες χώρες. Ε, όταν έχουμε διποτε δραστηριότητε, θα πρέπει να κατανοούμε τη φορολογική νομοθεσία στην εκάστοτε χώρα και είναι πολύ περίπλοκες. Γι' αυτό έχουμε και φοροτεχνικούς και έχουμε και συμβούλους για να κατανοήσουμε, για να συμμορφωθούμε προς τις υποδείξεις και την νομοθεσία της κάθε χώρας. Σε σχέση με το φορολογικό μας τμήμα στην Ευρώπη έχουμε οκτώ ε, υπαλλήλους που ασχολούνται με όλη την Ευρώπη και με κάποιες άλλες δικαιωτικές περιφέρειες και σε όλο τον κόσμο είναι καμιά πενινταριά στην Apple που εργάζονται ακριβώς στο φορολογικό τμήμα δεν είναι για την φορολογική βελτιστοποίηση, δηλαδή να πληρώνουμε λιγότερο, να έχουμε φορολογικά πλεονεκτήματα. Απλώς είναι για να δίνουν συμβουλές για τις αστεριότητές μας και να επεκτηνόμαστε παγκοσμίω και να βεβαιωνόμαστε ότι συμμορφωνόμαστε προς τη φορολογική νομοθεσία της κάθε χώρας. Σε ό,τι αφορά τώρα την Ιταλία συγκεκριμένα, Έχουμε λογιστικούς φορολογικούς ελέγχους και στην Ιταλία όπως και αλλού από καιρού εις καιρό και πρόσφατα σε, μια, σε ένα τέτοιο φορολογικό έλεγχο διαφωνήσαμε με την Ιταλική εφορία ε, σε σχέση με την εφαρμογή του νόμου και ως αποτέλεσμα αυτής της διαφωνίας ε, η Ιταλική εφορία ε, επέβαλε ε, έτσι, ένα φόρο κατά αποκοπή και εμείς το πληρώσαμε. Από την ΙΕΝΕΦ e ο χονό. Ποιον θα ρωτήσετε. Μόνο την Google εγώ. Δύο ερωτήσεις έχω. Κύριε Κοέν, ο πρόεδρο σα, κύριο συνεχίζει να μα λέει ότι σέβεται τον νόμο παντού και τον τηρεί η Google που έχει business. Ο τύπο όμω δημοσιεύει ε, άλλα πράγματα. Εκατοντάδες εκατομμύρια χάνουν οι ευρωπαϊκέ χώρες από ε, τα τεχνάσματά σα και τα τρίκ. Και η Google σύμφωνα με την ε, διαφήμιση που κάνετε είναι μια επιχείρηση πραγματικά υποδειγματική από πλευρά συμπεριφορά πολίτου. Φορολογικά όμω, έχετε ένα σύνταγμα δικηγόρων και συμβούλων για να ε, παρακάμπτετε τη φορολογική νομοθεσία. Και επίσης έχετε δωρεάν και το επαλαμβάνω εθνικές υποδομές στις οποίες ε, αξιοποιείτε που πληρώνουν οι πολίτες και επιχειρήσεις. Η καινοτομία και η νέα ε, οικονομία πρέπει να είναι γενναιόδορη. Εσείς είστε εγωιστές στο επιχειρηματικό σας μοντέλο και φακελώνετε και τους, πολίτες, ε, τους πελάτες σας ε, για αποκλειστικά προνόμια δικά σας για τις εταιρείες σας. Σήμερα το Βέλγιο και το Ηνωμένο Βασίλειο είναι θύματα της καταχρηστικής φορολογικής σας τακτικής και σας δούνε τα ρέστα. Για τη Γαλλία μπορείτε να μας πείτε που βρίσκεται η διαδικασία φορολογικού ελέγχου που σας επιβάλλει ε, το κράτος. 1,6 δις ακούμε ε, ε, ότι είναι φοροσετεριών εταιριών. ποια είναι τα διαστήματα που ελέγχθηκαν και που ελέγχονται. Για το μέλλον, θα σεβαστείτε την έκθεση αναχώρα. Ε, ακόμα και αν δεν είναι υποχρέωση από τον νόμο εθελοντικά. Υπάρχει μια ομάδα εργασίας ad hoc θα συνεργαστείτε ε, με τις ομάδες αυτές για την ε, επιθετική βελτιστοποίηση ε, τη φορολογική και την καταπολέμησή τους. Ευχαριστώ κύριο Σκόεν. Ευχαριστώ. Σε ό,τι αφορά τον ισχυρισμό ότι χάνει λεφτά η Ευρώπη, θέλω να το διευκρινίσω αυτό. Σύμφωνα με το Διεθνές Φορολογικό Δίκαιο, εμείς πληρώνουμε σε όλες τις χώρες που δραστηριοποιούμαστε τους φόρους μας. Οι φόροι που πληρώνουμε είναι αντικείμενο λογιστικού ελέγχου, φορολογικού και καμιά φορά προσαρμογή, όπω είδαμε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Υπάρχουν και σε άλλε χώρε διαδικασίε που τρέχουν, που ακούμε και περιγράφονται και δεν νομίζω ότι θα ήταν σκόπιμο να σχολιάσω ε, ανοιχτέ περιπτώσεις. Μόλις λυθούν θα επικοινωνήσουμε εμείς ε, μέσω των επισήμων διάβλων και των ε, λογαριασμών μα. Ε, το θέμα αυτό έχει να κάνει με τις ευρωπαϊκές υποδομές. εμείς είμαστε μαζικοί επενδυτές ευρωπαϊκές ε, ε, ε, υποδομές, δεν τις χρησιμοποιούμε απλώς, τις κατασκευάζουμε κιόλας. Και αν δείτε τις επενδυτικές μας δαπάνες είναι δισεκατομμύρια ευρώ. προηγουμένως σας απάντησα για τα υπόλοιπα που ρωτήσατε. Ε, για την αναφορά αναχώρα. Το 2017 αρχίζουν να το εφαρμόζουν διάφορες χώρες, αργότερα όλες οι εταιρείε και σίγουρα και εμείς θα συμμορφωθούμε με αυτό. Αυτό οδηγήσει σε μεγαλύτερη διαφάνεια και καλύτερη κατανόηση για το πώς ε, εφαρμόζονται οι φορολογικοί κανόνες στις πολυεθνικές. Αυτό θα ήταν ένα πάρα πολύ θετικό βήμα. Σας ευχαριστώ. Έχετε συμπληρωματική ερώτηση, Μπερνάρ. Ζητώ συγγνώμη. Δεν απάντησε ο κύριο Κοέν για το τζίρο και για τα κέρδη ε, που πραγματοποίησαν στη Γαλλία αυτή ε, που γίνεται ο έλεγχο. Θα ήθελα συγκεκριμένη απάντηση με στοιχεία, παρακαλώ. Αριθμητικά. Δεν τα έχω όλα αυτά τα τελευταία γαλλικά στοιχεία. Μπορώ να σας πω όμως ότι το 2013 ε, είχαμε 22 εκατομμύρια ε, κέρδη και προφόρου και πληρώσαμε φόρο 7,8 19,9 το 2013 και πληρώσαμε φόρο 5 εκατομμύρια ευρώ για την περίοδο αυτή. Πολύ ωραία και σας ευχαριστώ. Από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, ο Μπράιν Hayes. Εσείς σε ποιον θέλετε να ρωτήσετε και τους δύο. Μια γενική ερώτηση και προς τους δύο. Πρόεδρε, και μια ειδική ερώτηση στην Apple. Και τις δύο εταιρείε. θέλω να ρωτήσω για το Knowledge Box που είναι ε, ε, μια νέα δράση, φορολογική προσφορά σε διάφορα κράτη-μέλη. Το χρησιμοποιείτε και η μια εταιρεία και η άλλη για να μειωθεί ο φόρος που σας ζητούν κάποιες χώρες και να επενδύσετε στην έρευνα και την ε, ανάπτυξη. Γιατί από τη διαδικασία BEPS τώρα ε, νέες συνθήκες χρησιμοποιείτε λοιπόν αυτή τη νέα δομή, το knowledge box στο Ηνωμένο Βασίλειο και από ό,τι φαίνεται και στις κάτω χώρες ισχύει αυτό. Και συγκεκριμένη ερώτηση προς την Apple, Πρόεδρε. Και χαίρομαι για το γεγονός ότι στην Ιρλανδία έχουν 5.500 ε, άμεσα εργαζομένους και 18 έμεσα. Ε, θέλω να ρωτήσω κάτι που ρώτησε και ο Φάμπιο μαζί προηγουμένως. Ως Apple θεωρείτε ότι έχετε άδικη μεταχείριση, άνηση μεταχείριση για την έρευνα που γίνεται για τον ανταγωνισμό και τι πιστεύετε για την έρευνα αυτή ή άλλες έρευνες αντίστοιχες από αρχές ανταγωνισμού στις Ηνωμένες και αλλού. Και επίσης θέλω να σας ρωτήσω, κάποιος είπε πρόσφατα ότι ανεξαρτήτως το αποτελέσματος θα παραμείνει Apple στην Ιρλανδία, είναι 40 χρόνια τώρα και εδρεύει εκεί και ε, θέλει να εδρεωθεί. Ό,τι και να γίνει, ό,τι και να βγει θα παραμείνει. Αν συμβεί κάτι τέτοιο και δεν έχω κανένα λόγο να τον φυσβητώ, πώς θα παραμείνετε στην Ιρλανδία δηλαδή και μπορείτε να ε, επεκταθείτε στην απάντησή σας με τα στοιχεία που θα δώσει στην Επιτροπή. Να αρχίσουμε με την για αυτό το knowledge box ε, δεν χρησιμοποιούμε τίποτα σχετικό μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. <laughs> So, Apple. Apple. Ούτε εμεί χρησιμοποιούμε τέτοια ξεχωριστά φορολογικά καθεστώτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε για τα πνευματικά δικαιώματα, είτε για την έρευνα και ανάπτυξη των Knowledge Box. Ε, και ξαναλέμε, όσο επιτοπλίστων, διεξάγουμε τι δραστηριότητε μα ε, στη ΣΥΠΑ και γι' αυτό εκεί επικεντρώνουμε την προσοχή μα, ε, διότι εκεί έχουμε όλες τι δραστηριότητε έρευνα και ανάπτυξη. Φυσικά, βάσει και τη μελλοντική νομοθεσία μπορεί και να επεκταθούμε, αλλά ω επιτοπλίστων στην Αμερική. Ε, θέλω να απαντήσω στις υπόλοιπες ερωτήσεις. Αν ε, θεωρούμε ότι στα πλαίσια κρατικών προμηθειών υπάρχει άνεση μεταχείριση. Δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε τι ισχύει για τις υπόλοιπες εταιρείες. Εμείς ε, έχουμε πλήρη συμμόρφωση. Θεωρούμε ότι ό,τι χρωστούσαμε το πληρώσαμε μέχρι τελευταία δεκάρα στην Ιρλανδία και δεν ε, τίθεται ζήτημα κρατικών προμηθειών. Νομίζω ότι θα αποδειχθεί ε, το ορθό των ε, δηλώσεών μας και πιστεύω θα μας στηρίξει και η Ιρλανδική κυβέρνηση. Γιατί είπα, δεν είμαι σε θέση εγώ να παραβάλω δύο διαφορετικά συστήματα. Για το, την παρουσία μας στην Ιρλανδία και τις επενδύσεις στην Ιρλανδία έχουμε δέσμευση, στενή σχέση και με την Ιρλανδία και με την Ευρώπη και το αποδεικνύουμε αυτό. Κάθε μέρα, ε, είδατε τις ε, πρόσφατες δηλώσεις στη Δανία και στην Ιρλανδία, ανοίγουμε κέντρα μασικών ε, δεδομένων, επεκτηνόμαστε. Φυσικά θα παραμείνουμε στην Ευρώπη. Ο Μπράιν έχει κοκκινήσει. for Η Ελίζα Φερίρα από τους σοσιαλιστές. Μία ερώτηση προς την Apple και μετά Google. Θυμάστε την έρευνα 2013 από τη Γερουσία τον είπα. Ο κύριος Τιμ Κουκ που εκπροσωπούσε την εταιρεία σας ε, έδωσε κάποιες απαντήσεις συγκεκριμένως όταν ο Κάρλ Λέβιν, ο γερουσιαστής, κατηγόρησε την Apple ότι έχει τρεις ε, offshore εταιρείε και αυτές οι οντότητες ε, λαμβάνουν σε έσοδα δεκάδες ε, δισεκατομμύρια όμως δεν έχουν φορολογική έδρα. Και τι απάντησε η εταιρεία σας, ναι κύριε, δεν έχουν φορολογική έδρα ούτε η μία ούτε η άλλη. και για τη σχέση είπα σας κατηγόρησαν ότι ε, είχατε ε, διαπραγματευτεί ένα συντελεστή 2% κάτω από τον ε, κανονικό φορολογικό συντελεστή του 12,5%. Και όταν ερωτήθη ο Τιμ Κουκ είπε ότι αυτός ο φορολογικός συντελεστής είναι για προϊόντα που πολλούμε εκτός και όχι εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. στο τζίρο σας το 55% των εσόδων ε, ε, έρχονται από χώρες εκτός των ΗΠΑ. Μήπως να πληρώνατε και φόρους αφού έχετε τις ε, δραστηριότητες στην, στην Ευρώπη. Μετά, είπατε ότι όπως και όλοι οι υπόλοιποι ε, με την νομοθεσία. Εσείς πώς αντιλαμβάνεστε ακριβώς την κοινωνική εταιρική ευθύνη Έχετε τέτοια στρατηγική για το εργατικό δίκαιο, για την υγεία, για το προσωπικό και δηλαδή εκμεταλλεύεστε το έπακρον όλα τα παραθυράκια. Όμως μας εμπνέει αυτό που κάνετε στο ρόλο του συνομοθέτη. Ωραία. Apple. Για τη μη φορολογική έδρα, αυτό που είπατε ότι οι θηγατρικές δεν έχουν φορολογική έντρα. Στην Ιρλανδία ε, είναι εκεί οι εταιρείε, αλλά τις διαχειρίζονται η όλες Όλες οι δραστηριότητες για τα πραγματικά δικαιώματα ε, είναι στη ΣΥΠΑ. Η στρατηγική για το μάρκετινγκ, όλες, οι ε, κατευθυντήριες γραμμές προέρχονται από τη ΣΥΠΑ. Αυτό απορρέει από την Ιρλανδική νομοθεσία. Προβλέπεται να υπάρχουν εταιρείε που δεν έχουν φορολογική έδρα. Ε, το αντίστοιχο σημαίνει και ΣΥΠΑ. Από Ιρλανδική σκοπιά ή Αμερικανική τότε δεν είχαν φορολογική έδρα. Okay. Μας ρωτήσατε για την κοινωνική εταιρική ευθύνη. Και αν ε, σεβόμαστε το εργατικό δίκαιο, την νομοθεσία για την υγεία, απολύτως συμμορφωνόμαστε όπου και αν διεξάγουμε τις ε, δραστηριότητές μας, ε, καταβάλουμε φόρους όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Και είμαστε περήφανοι για αυτό που προσφέρουμε στην Ευρώπη. 14.000 εργαζόμενους έχουμε. Ε, έχουμε ε, και την καινοτομία σε μικρές ψηφιακές επιχειρήσεις ε, που είναι σαν δορυφόροι της Google και από εκεί προκύπτει μεγάλη καινοτομία και πολλές θέσεις εργασίας. Αλλά ξέρουμε ότι ούτως ή άλλως τα ψηφιακά μέσα έχουν αναπτυχθεί πάρα πολύ. Άλλωστε γνωρίζουμε και την εξέλιξη που είχε ε, ξεκινώντας από τις ΗΠΑ ε, το ε, διαδίκτυο. Ωστόσο, δημιουργήθηκαν μόνο τις, τα τελευταία δύο χρόνια 200.000 θέσεις εργασίας και 11 δις λίρες το, ο τζίρος μας. Ναι, αλλά δεν θεωρείτε λέει κυρία Φεραίρα ότι το γεγονός ότι να πληρώνετε 2 ή έστω 3% επί των κερδών σας δεν είναι ε, λογικό τη στιγμή που ένας απλό ε, πολίτης ή κάποιος άλλος θα πληρώσει 30% ε, και συμβάλλουν περισσότερο τελικά στον προϋπολογισμό. Είναι καλό για τη φήμη σας αυτό. Ε, μα τέτοιου είδους ε, ε, στοιχεία θέλουμε να συζητήσουμε γιατί δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα φορολογικέ μα μας υποχρεώσεις στου διεθνεί κανόνε που ισχύουν. Θέλω να συμμετάσχω στη συζήτηση για να υπάρξει καλύτερη κατανόηση <clears throat> για τους φορολογικούς κανόνες και να συμβάλλω και στη εργασία σας. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό για να διαπιστώσουμε πρέπει ή δεν πρέπει να αλλάξουν οι κανόνες. Πρόεδρος, μα εμείς είμαστε οι συνομοθέτες, αλλά δυστυχώς στα φορολογικά ζητήματα ε, νομοθετούν τα εθνικά κοινοβούλια. Ε, δυστυχώς και όχι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οπότε βουλευτές σαν και εμάς θα αποφασίσουν. Ε, οι πολίτες μπορούν να έχουν την άποψή τους, αλλά εμείς αποφασίζουμε και το τονίζω. Επανειλημμένα θέσαμε αυτά τα ερωτήματα στους προσκεκλημένους μας για τις επιχειρήσεις αν είναι παράνομη ή νόμιμη η δραστηριότητα, αν είναι δίκαιο ή όχι. Ε, εμείς αποφασίζουμε, το τονίζω. Πάλι τα... Ευχαριστώ Πρόεδρε. Τρεις σύντομε ερωτήσει για την Google και για την Google μόνο. Ναι, μόνο για την Google. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση να έρθουμε στο Google Netherlands και μερικά μέλη από το κόμμα μου ε, ε, θέλουν πάρα πολύ να δούμε πώς λειτουργεί αυτή η θηρίδα εταιρεία. Ένα γραμματοκιβώτιο έχετε εκεί πέρα. Ε, έχετε και στο Άμστερνταμ λοιπόν μια τέτοια εταιρεία για να μπορείτε να ε, πληρώνετε φόρους ή να μην πληρώνετε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι το λέτε. Έτσι. Αυτό χωλένει έτσι και αλλιώς από μόνο του. Γιατί διαλέξατε αυτή τη θηρίδα λοιπόν στο Άμστερνταμ τη συγκεκριμένη. Δεν θα μπορούσε να είναι κάπου αλλού. Υπήρχε κανένας ιδιαίτερος λόγος στο Άμστερνταμ. The specifics of the ε, ε, συγκεκριμένα και οι κανόνες για το πώς ε, αυτό επελέγει με, με ξεπερνάει. Δηλαδή ήταν πριν τη δική μου εποχή, ήταν 40 χρόνια πριν, δεν είχα καν γεννηθεί για να καταλάβετε. Το βασικό, της ερώτησης αυτής, ο βασικός κορμός γιατί χρησιμοποιείται μια δομή και αν, αν ήταν κάπου αλλού θα είχε διαφορά, όχι. Ε, ή θα αποφεύγαμε κάποιες ευρωπαϊκές ή αμερικανικές υποχρεώσεις για την Αμερική ναι γιατί δεν επαναπατρίζουμε κέρδη για την Ευρώπη όχι θα μπορούσε λοιπόν να είναι οποιαδήποτε χώρα και για να το διατρανώσω και πάλι δεν ε, ε, αλλάζει καθόλου τις υποχρεώσεις που έχουμε στην Ευρώπη στις δικαιοδοτικές επικράτες Πάουλ, η Ολλανδική Βουλή θέλει να βεβαιωθεί ότι πληρώνεται φόρους στην Ολλανδία. Υπάρχει μια συμφωνία με την εφορία της ε, ε χώρας. Ε, θέλετε να το συζητήσετε αυτό με την Ολλανδική Βουλή. Δεν ξέρω εγώ να έχουμε συμφωνία με την Ολλανδική Εφορία. Χρησιμοποιούμε τις δομές που υπάρχουν και τους κανόνες που ισχύουν για όλες τις πολυεθνικές εταιρείες που έχουν ε, αντίστοιχε δομέ. Άλλο ρώτησα λέει. Υπάρχει ένα tax ruling με την ε, Ολλανδική εφορία. Είστε πρόθυμοι να έρθετε να τα συζητήσετε αυτά με την Ολλανδική Βουλή. Δεν ξέρω για ποιο πράγμα μιλάτε και για ποια συμφωνία. Όπως σας είπα, ε, αυτό έγινε πριν γεννηθώ, πριν έρθει η Google. Το χρησιμοποιούν ευρέως πολλές πολυεθνικές αμερικανικές στην Ευρώπη. Ωραία. Να επανέλθω λοιπόν από άλλη σκοπιά. Στην Google έχετε κώδικα δεοντολογίας, έτσι. Και είναι πολύ απλός και δεν θα πρέπει να έχετε ε, σύγκρουση συμφερόντων και αν ε, κάτι ε, βγει στον τύπο που σας ενοχλεί εσάς ή την Google. Λοιπόν, από αυτά που συζητάμε τώρα και που λέτε εδώ, θεωρείτε ότι σας ενοχλεί κάτι. Δηλαδή, τι εννοείτε, ότι δεν θα έπρεπε να είμαι παρόν. Με καλέσατε, όπως και το συνάδελφο τον Νοέμβριο, για συμμετέχουμε σε μια επικοδομητική συζήτηση για το πώς μπορούν να αλλάξουν οι κανόνες. Γι' αυτό ήρθαμε και χαιρόμαστε να συμμετέχουμε στη συζήτηση αυτή. Υπάρχουν θέματα ουσίας που προσπάθησα να σας εξηγήσω, να βοηθήσω στις εργασίες της Επιτροπής σας και είμαι βέβαιος ότι οι συνάδελφοι ε, θα ε, χαρούν για το γεγονός ότι το πράττω εξ ονόματός τους. Δηλαδή ποιον εκθέτει ε, κάμερ δηλαδή ε, η Ολλανδική Βουλή πρέπει να καλέσει την Google. Ε, πάντως έρχονται, οπότε τους ε, καλούμε. ECR, η κυρία ε, Γόνολε, ποιον θέλετε να ρωτήσετε από τους δύο. Ευχαριστώ, Google. Πόσο εταιρικό φόρο πληρώσατε πέρσι? Και σε ποια χώρα. Προσπάθησα <laughs> να το ψάξω στο Google, αλλά απάντηση δεν βρήκα. Η αποστολή σας είναι, και παραθέτω αυτά που λέτε στην ιστοσελίδα σας, να διευκολύνετε πρόσβαση στις πληροφορίες για ε, ολόκληρο τον κόσμο. Τα καταφέρνετε, πιστεύετε. Η εταιρική κοινωνική ευθύνη που έχετε, όπως την εκφράζετε σε μία δήλωση, προβλέπει ότι υπάρχει μεγαλύτερη συνειδητοποίηση των φιλανθρωπικών εταιρικών δραστηριοτήτων. Το 2014 πληρώσατε σχεδόν 12 δις σε εντελώς αδιαφανείς εταιρείες στις Βερμούδες που δεν έχουν σχέση με τις επιχειρηματικές σας δραστηριότητες. Αυτή είναι νέα εκδοχή της επιχειρηματικής φιλανθρωπίας και πριν από έξι χρόνια η Google αποφάσισε να αποσυρθεί από την Κίνα. Και τότε σκέφτηκα. Μα καταπληκτική εταιρεία. Τώρα ξαναπροσλαμβάνεται στην Κίνα, διαβάζουμε σε εφημερίδες. Πότε θα ξαναγίνεται η παλιά, η καλή Google. Ευχαριστώ. Κοέν. Για τους φόρους που πληρώσαμε πέρσι. Ε, στις αιτήσεις λογαριασμούς μας υπάρχουν τα πόσα και σας τα δίνω. 3,3 δις πληρώσαμε, αμερικανικά δολάρια, έτσι, για το 2015, 2,6 δις, ε, ε, ε, ομοσπονδιακοί φόροι. 706 εκατομμύρια δολάρια είναι το σύνολο των φόρων. Ακόμη δεν έχουμε ολοκληρώσει λογαριασμού ε, για τι ευρωπαϊκέ χώρε. Ε, μπορώ να σα πω όμω ότι πληρώσαμε σε διάφορε ε, χώρε Ευρωπαϊκή Ένωση το 2014. Όλα αυτά είναι δημόσιε πληροφορίε, δημόσια προσβάσιμε πληροφορίε και ελπίζω το, η μηχανή αναζήτηση του Google να λειτουργεί καλά και να τα βρίσκεται αυτά, αλλά πάντω είναι διαθέσιμε οι πληροφορίε. για την επιχείρηση στις Βερμούδες, ε, την οντότητα στις Βερμούδες, ε, νομίζω ότι εξήγησα ότι αυτό δεν επηρεάζει είναι τους φόρους που πληρώνουμε στην Ευρώπη και σχετίζεται με ιδιαιτερότητα του Αμερικανικού Ομοσπονδιακού Φορολογικού Συστήματος αυτό το διπλό Ιρλανδικό σάντουιτς ε, ε, εκπνέει το 2020 βάσει των κατευθυντηρίων γραμμών του ΩΣΑ και αλλάζουν οι κανόνες στην Ιρλανδία μετά από αυτές τις κατευθυντήριες του ΟΣΕ. Για τις ερωτήσεις για την Κίνα. Ειδικό δεν είμαι για αυτή την περιοχή γιατί ε, έφτασα στην Google όταν έφυγε από την Κίνα. Εμείς έχουμε αυτό το pullback που λέμε, η απόσυρση από την ε, Κίνα έγινε ε, λόγω της λογοκρισίας ε, των αποτελεσμάτων αναζήτησης από την κινέζικη κυβέρνηση. Και από ό,τι ξέρω εξακολουθεί να ισχύει αυτό. Ευχαριστούμε. Ο Παύλο ο Σάλβα. Τώρα θέλεις να μιλήσεις Παύλο. Για ποιον η ερώτηση. Θα τα πω ισπανικά. Ε, μια για την Apple και μια γενική. Εσείς είπατε ότι δεν δημοσιοποιείται ε, το πόσους φόρους πληρώνετε σε κάθε χώρα. Για ποιο λόγο υπάρχει κανένας λόγος που δεν τα δημοσιεύετε αυτά τα στοιχεία και δεν πιστεύετε ότι μια εταιρεία του κύρους ε, το οποίο χαίρει η Apple και μάλιστα όχι μόνο ο κύρος και θαυμασμό νιώθει ο κόσμος. Ε, θα ήταν σκόπιμο να τα δημοσιοποιεί για να μην βλάψει την εικόνα της σε κάθε χώρα. Αλλιώ δίνετε την εντύπωση ότι κάτι θέλετε να κρύψετε. Ενώ δεν νομίζω καθόλου ότι είναι η πρόθεσή σα. Είμαι βέβαιο γι' αυτό. Και μια γενική ερώτηση σε όλου. Πήραμε κάποια μέτρα, κάναμε κάποια βήματα. Θέλω να σα ρωτήσω, εσεί έχετε καμιά πρόταση να κάνετε σχετικά τι θα μπορούσαμε να προτείνουμε εμείς από την Επιτροπή Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Η Apple. Oh, για την δημοσιοποίηση των φορών πληρώνουμε. Το βασικό για μας είναι ότι λειτουργούμε σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον και βασικά Πιστεύουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για μας και όχι μόνο για οποιονδήποτε λειτουργεί σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Θέλουμε ισότιμους όρους ανταγωνισμού όταν ε, δημοσιεύουμε. Οπότε όταν όλοι πρέπει να το κάνουν και γίνεται με συνέπεια σε όλες τις χώρες, με τα χαρά να το κάνουμε κι εμείς. Μέχρι τότε όμω είναι εμπιστευτικέ πληροφορίε των προλογουμένων προστατευόμενο αυτό το δικαίωμα και από την νομοθεσία. Όταν προβλεφθεί από τον νόμο θα το κάνουμε και εμείς. Με μεγάλη χαρά. Τζούλια, θέλεις να ε, ε, ε, σχολιάσεις το θέμα των προτάσεων. Είναι λίγο νωρίς για προτάσεις, αλλά άμα θες... Ναι, όπως είπες και εσύ, για αυτά που συζητούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα Ε, δεν έχουμε ακόμη μη θέση, αλλά οι πολυμερείς συζητήσεις και αυτές που γίνονται στην Ευρώπη είναι σημαντικές όταν βλέπουμε τα όσα συμβαίνουν τώρα για την ε, φορολογική μεταρρύθμιση σε ολόκληρο τον κόσμο και για τη συνεπή εφαρμογή των νέων διατάξεων. Όταν βλέπετε αυτούς τους κανόνες, ε, σε όλους, φαίνεται ότι πρέπει να δούμε μια διαφοροποίηση ως προς την εφαρμογή των νέων κανόνων. Αυτή η πολυπλευρή προσέγγιση ε, είναι αυτό που προτείνω και η συνεπή εφαρμογή από τις επιχειρήσεις. Αυτό σας πρότεινα. Ωραία. Ευχαριστώ. Τελειώσαμε με την ανταλλαγή πληροφοριών για το πρώτο πάνελ. Ευχαριστούμε σε εκπροσώπους Google και Apple. Διακόπτουμε για ένα λεπτό ώστε να έρθουν οι εκπρόσωποι McDonald's και η και Ήσασταν στο κοινό να, μέχρι να έρθουν να σας αντικαταστήσουν. Δεν σας ε, αποπέμπω κύριε Κοέν και κυρίες μου. Αν θέλετε να μείνετε.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 Bien, Τέρμα το διάλειμμα. Nous reprenons Ξαναρχίζουμε λοιπόν τις εργασίες μας και τώρα θα ξεκινήσει το δεύτερο πάνελ. Και καλωσορίζω τον κύριο Σόρεν Άμσεν, ο οποίος ε, είναι ε, ο εκτελεστικός διευθυντής της IKEA και την κυρία Ειρήν Γέιτς, η οποία είναι αντιπρόεδρος, υπεύθυνη ε, για θέματα εταιρικού, ε, εταιρικής φορολογίας ε, του McDonald's. Και είναι, είναι παρόν επίσης και ο υπεύθυνο επικοινωνίας του IKEA. Όχι, συγγνώμη, συγγνώμη. Όχι, ναι, δεν είστε, δεν είστε στην McDonald's, τουλάχιστον όχι ακόμα, τουλάχιστον όχι ακόμα. Ίσως μετά από το πέρας αυτής της ε, συνεδριάσεως να αποφασίσετε να αλλάξετε στρατόπεδο. Πολύ ωραία. Ε, ακούσατε λοιπόν το πρώτο τμήμα ε, ε, γνωρίζετε επομένως τους κανόνες ε, του παιχνιδιού και τον χρόνο παρέμβασης. Έχετε πέντε λεπτά έτσι ώστε να κάνετε την αρχική σας παρουσίαση, δηλαδή την στρατηγική, τη φορολογική της, του ομίλου σας και μετά θα δώσουμε τα, τον λόγο στα μέλη σύμφωνα με χρονοθυρίδες αυστηρά πέντε ετών, λεπτών συγγνώμη, ε, και θα έχουν τη δυνατότητα λοιπόν ε, να ε, να, θα έχετε τη δυνατότητα να απαντήσετε και θα έχετε πάλι δύο και ένα λεπτά, τρία λεπτά λοιπόν για να απαντήσετε. Έχετε το λόγο για πέντε λεπτά. Thank you very much. Mr. Chairman, Κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είμαι ο Σόραν Χάνσενε και είμαι Διευθύνων σύμβουλο του ε, ομίλου IKEA. Ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε και μου δώσατε τη δυνατότητα να συμμετάσχω σε αυτήν την ε, συνεδρίαση τη ειδική ε, επιτροπή σα για θέματα τα οποία σχετίζονται με το CCCTB και το BEPS και άλλα φορολογικά ζητήματα. Στο τέλο τη δεκαετία του 80, αρχέ του 90 ήταν πάρα πολύ δύσκολο να επεκταθεί αναφερθεί στην, ε, ε, συγγνώμη, τέλη δεκαετία του 70 και αρχέ τη δεκαετία του 80 ήταν πάρα πολύ δύσκολο να ε, διευρύνει κανείς την παρουσία του στην Ευρώπη. Η εξέλιξη όμως της αγοράς, στην αγορά ήταν ε, και η διεύρυνση της βάσης μας ήταν απολύτως απαραίτητη έτσι ώστε να βελτιώσουμε την παρουσία μας στην Ευρώπη. Ε, παρακολουθήσαμε με πολύ μεγάλη προσοχή ναι, τη συζήτηση που γίνεται για την ε, φορολογία των επιχειρήσεων ε, τα τελευταία χρόνια και παρακολουθούμε και στενά όλες τις επικρίσεις που ακούγονται σχετικά με τον όμιλο IKEA. Βεβαίως εμείς πιστεύουμε ότι πάντα μπορεί κάποιος να μάθει κάτι μέσα από τη συζήτηση. Ο όμιλος IKEA πληρώνει τους φόρους της οπουδήποτε λειτουργεί και είναι εγκατεστημένη Οι, διαφορετι... οι διάφορες εταιρείες μας βεβαίως πληρώνουν διαφορετικό... Ε, διαφορετικούς ε, φόρους και όσον αφορά την ιδιοκτησία, τα κέρδη ή άλλου είδους ε, φορολογήσεις. Η... Το ποσοστό της φορολόγησης και ο τρόπος καθορίζεται από τον νομοθέτη της εκάστοτε δικαιοδοσίας. Εμείς συμμορφούμαστε με τις... συμμορφωνόμαστε με τα όσα αναφέρει ο νομοθέτης. Θεωρούμε ότι μια υγιής ε, επιχείρηση είναι σημαντικός μοχλός ανάπτυξης ε, της ε, επιχείρησης. Και πιστεύουμε επίσης ότι μια σαφής φορολογική νομοθεσία μπορεί να δώσει συγκεκριμένες λύσεις χωρίς να βαραίνει, χωρίς να βαραίνει γραφειοκρατικά την, τις επιχειρήσεις. Ε, υπάρχουν πολλά ζητήματα κύριε Πρόεδρε τα οποία ε, σχετίζονται με παρανοήσεις όσον αφορά το σύστημα franchise ε, της, του, του, του ομίλου IKEA. Η, IKEA δεν είναι μία εταιρεία ή ένας όμιλος εταιριών. Είναι διάφορες εταιρείες. Η Inter IKEA Group είναι αυτή η οποία κατέχει τις άδειες franchise τις οποίες δίνει στις επιμέρους εταιρείες. Και τα μέλη της ε, IKEA Group ε, λειτουργούν κάτω από την ομπρέλα του brand name της ε, IKEA. Από το 1993 υπάρχει και η έννοια του franchisor του franchisor της, της IKEA με συγκεκριμένη παροχή συμβουλών κτλ. Εμείς ας πούμε στην ε, ε, Ολλανδία είχαμε μια συμφωνία franchise ε, με χίλιους, με χίλιους εργαζόμενους. Η κάθε συγκεκριμένη franchise συμφωνία αφορά τη συγκεκριμένη χώρα. Έχουμε 13 τέτοιες συμφωνίες αυτή τη στιγμή και ο μόνος, ε, ε, ε, η μόνη ομάδα η οποία μπορεί να θεωρηθεί ομάδα IKEA είναι αυτή η οποία εντάσσεται μέσα στο σύστημα Inter IKEA έχοντας πάνω από 13 franchisees στην δικαιοδοσία του όλοι οι franchisees της IKEA πληρώνουν 3% ε, κόστος ε, franchising ε, στο Inter IKEA Group και αυτά τα χρήματα καταβάλλονται, έχουν σαν τελικό αποδέκτη την εταιρεία που έχει έδρα στην Ολλανδία. Είναι γεγονός ε, ότι η επιχειρησιακή μας στρατηγική πολλές φορές ε, θεωρείται από πολλούς ιδιαίτερα περίπλοκη. Αλλά ε, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι μέχρι τώρα έχει λειτουργήσει καλά. Έστω και αν αναγνωρίζουμε ότι παρόλα αυτά υπάρχουν τομείς οι οποίοι χρήζουν περαιτέρω βελτιώσεων. Εμείς ακολουθούμε την αρχή της διαφάνειας και μάλιστα πέρα και παραπάνω από τις υποχρεώσεις που καθορίζει η νομοθεσία Έχουμε ε, δημοσιοποιημένες ε, εκθέσεις ε, στις περισσότερες χώρες. Εμείς μπορεί να εξακολουθούμε να κάνουμε λάθη, είναι βέβαιο αυτό, αλλά σας διαβεβαιώ ότι εμείς θα συνεχίσουμε την προσπάθειά μας για απλούστευση των διαδικασιών που οπωσδήποτε θα έχουν εν τέλει μεγαλύτερη, σαν αποτέλεσμα μεγαλύτερη διαφάνεια και μεγαλύτερη σαφήνεια των φορολογικών Όσον αφορά τώρα την BEPS ε και την CCCTB θεωρούμε ότι πρόκειται για αρχές οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν στην απλούστευση και εν τέλει στη βελτίωση ε, του, ε, της καταστάσεως. Αυτά μέχρι τώρα, τον διακόπτει ο Πρόεδρος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και έχετε τον λόγο εσείς κυρία Γέιτσε. Καλό απόγευμα. Είμαι υπεύθυνη για την φορολογία, για, την ε, φορολογία της επιχείρησης McDonald's. Και την προηγούμενη χρονιά είχαμε ε, έρθει ενώπιό σας έτσι ώστε να συζητήσουμε τις προτάσεις BEPS και CCCTB. Ε, είναι πολύ καλή ευκαιρία που μας δίνεται και σήμερα έτσι ώστε να μπορέσουμε να πούμε δύο λόγια όσον αφορά την, την φορολογική διαφάνεια. Η εταιρεία McDonald's είναι απολύτως ε, αποφασισμένη να συμμορφώνεται με τα ε, συστήματα τα φορολογικά τα οποία ισχύουν σε κάθε χώρα στην οποία ε, δραστηριοποιείται είτε πρόκειται σε όλες τις περιπτώσεις πρέπει να σας πω ότι έχουμε τα τρία τέταρτα των εστιατορίων μας στην Ευρώπη βάσει του συστήματος franchising. Οι franchisees έχουν την την ε, δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν το όνομα, να χρησιμοποιήσουν επίσης κάποιες άλλες ε, εταιρικές ε, διαδικασίες και πληρώνουν ένα τέλος στην μητρική εταιρεία. Επίσης πρέπει να σας διαβεβαιώσω ότι η εταιρεία πληρώνει κάθε είδους φόρους σε κάθε δικαιοδοσία στην οποία είναι παρούσα. Είτε πρόκειται για φόρους επί των κερδών, είτε πρόκειται για φόρους ιδιοκτησίας κλπ. Ε, παραπάνω από 2,5 δις δολάρια πληρώνει η εταιρεία McDonald's καθαρά για φορολόγηση κερδών. Ε, αναφερόμαστε μονάχα στο καθαρό, ε, στους καθαρούς φόρους επί των κερδών που εφαρμόζονται, στις, στην κεντρική, που εφαρμόζονται επί του συνόλου της εταιρείας McDonald's. όσον αφορά το σύστημα των franchise, θεωρούμε ότι το 2000 2015 ε, η McDonald's μαζί με τους franchisees πλήρωσε πάνω από ένα δις ε, ε, ευρώ σε φόρους εταιρικούς. Όσον αφορά τώρα την δομή μας, την εταιρική μας δομή, Έχουμε ε, ένα σύστημα franchisees που χρησιμοποιούν ε, το λεγόμενο global brand ε, name. Έχουν, οι εταιρείε αυτές πληρώνουν πάντα royalties στην κεντρική εταιρεία, πράγμα που μας επιτρέπει να προχωρήσουμε σε πολιτικές ανάπτυξης και βελτιστοποίησης των προσφορών μας. Ε, οι μέθοδοι που χρησιμοποιούμε έχουν την σφραγίδα του ΩΣΑ και είναι αποδεκτές από τον ΩΣΑ. Όσον ε, αφορά τώρα στον ΠΕΠΣΕ και το CCCTB, εμείς καλωσορίζουμε αυτές τις νέες αρχές ε, γιατί θεωρούμε ότι με τον τρόπο αυτό θα υπάρχει μεγαλύτερη συνοχή στα φορολογικά συστήματα διεθνώς. Βεβαίως η ασφάλεια των, του δικαίου και η σαφή σαφήνεια των κανόνων είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ε, οι πολυεθνικές εταιρείες χρειάζονται ακόμα περισσότερο αυτήν την ασφάλεια των κανόνων έτσι ώστε να μπορέσουν να αναπτυχθούν η ανταλλαγή των πληροφοριών είναι πάρα πολύ σημαντική κατά την άποψή μας. Η McDonald's αναγνωρίζει ότι τα συστήματα ανταλλαγής πληροφοριών ε, πρέπει να βελτιωθούν. Θεωρεί ότι η αναφορά αναχώρα είναι μια θετική ε, εξέλιξη. Όσον αφορά τώρα ε, τον, ε, όσον αφορά την προσέγγιση αναχώρα, θεωρούμε ότι θα πρέπει τα οι φορολογικές μεταρρυθμίσεις να είναι τέτοιες έτσι ώστε να αρθούν τα, οι φραγμοί που υπάρχουν μεταξύ των χωρών έτσι ώστε να υπάρχει ταυτόχρονα μεγαλύτερη σαφήνεια, διαφάνεια και καθαρότητα της νομοθεσίας. Με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουν μεγάλες εταιρείες όπως η McDonald's να συνεχίσουν την ανάπτυξή τους ε, σε χώρες όπου ε, είναι ήδη παρούσα και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και οπουδήποτε στον κόσμο. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ κυρία μου. Θα δώσω το λόγο στον εισηγητή. Ευχαριστούμε και καλωσορίζω τους εκπροσώπους της και του McDonald's ε, με το Μακδόναλτ θα ήθελα να αρχίσω. Και μετά ε, την νοικία. Την περασμένη φορά που ήρθατε ήσασταν υπέρ της υποβολής εκθέσεων ανάχωρα αλλά κατά της ε, δημοσίευσης. Και όπως βλέπουμε το πακέτο για την ε, φοροαποφυγή από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα κατατεθεί και συγκεκριμένη πρόταση για τις εκθέσεις αναχώρα. Κύριε Γίτσε, είσαστε, εξακολουθείτε να είστε κατά τη δημοσίευση των εκθέσεων αναχώρα και αν ναι, γιατί. Επίσης, για το πακέτο αυτό της Επιτροπής, Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη φοροαποφυγή, πώς θα επηρεάσει αυτό το επιχειρηματικό ε, μοντέλο του McDonald's, αν εγκριθεί αυτό το πακέτο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα μας ενδιαφέρει να γνωρίζουμε ε, την απάντησή σας. Σας ευχαριστώ. Ναι, για τις εκθέσεις αναχώρα. Όπως και άλλες προσπάθειες εναρμόνισης, ε, είμαστε υπέρ της θέσπισης κοινού σετ κανόνε για την τεκμηρίωση, για την ε, μεταβίβαση ε, των κερδών καθώς και για τις εκθέσεις αναχώρα. Πιστεύω ότι δημοσιεύουμε ήδη πολύ σημαντικές λεπτομέρειες για τις δραστηριότητές μας και φορολογικές αρχές εποπτεύουν αυτά τα στοιχεία κατά τη συνεργασία μας με αυτές τις αρχές. Συμμετέχουμε και σε μια αξιολόγηση αντικτύπου για αυτό το ζήτημα και περιμένουμε τις, ε, τα αποτελέσματα και ε, θα συμμορφωθούμε με τις αποφάσεις, αν δηλαδή πρέπει να δημοσιεύουμε γενικά τις πληροφορίες ή να τις κοινοποιούμε μόνο στις φορολογικές αρχές. Σε σχέση με το πακέτο φοροαποφυγής, ε, ήθελα να πω ότι λειτουργούμε ε, αν χώρα και 75% των λειτουργιών μας, των δραστηριοτήτων μας, γίνονται από ανεξάρτητους επαγγελματίες. Ολιστική αποτίμηση δεν έχουμε κάνει εν μέρη διότι μένουν κάποια ερωτήματα αναπάντητα σε σχέση με το τι θα μπορούσε να συμβεί, αλλά θα θέλαμε να μάθουμε περισσότερα για ε, το πακέτο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να απαντήσουμε ε, αν απαιτείται αυτό. Ε, Επερώτηση. Δεν άκουσα κανένα επιχείρημα γιατί είσαστε κατά της δημοσίευση των πληροφοριών των εκθέσεων αναχώρα. Υποθέτω ότι αν το προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα αντιταχθείτε εσείς θα εφαρμόσετε τους κανόνες και θα είστε υπέρ. Ε, κατάλαβα καλά. Θέλω να σιγουρευτώ μόνο ότι κατάλαβα την απάντησή σας. Μικρόφωνο, δυστυχώς η ομιλήτρια μιλάει εκτός μικροφώνου. Ναι, συμμορφωνόμαστε με το φορολογικό δίκαιο και γενικότερα με την ενόμη της χώρας ε, όπου δραστηριοποιούμαστε, οπότε αν προβλέπετε αυτό, ναι, θα συμμορφωθούμε. Σε σχέση τώρα με τη θέση του Μακτόλα ε, για το γιατί προτιμούμε δηλαδή να μην είναι, δημοσιοποιούνται οι πληροφορίες. Υπάρχουν 150.000 άλλα ε, υποκαταστήματα που ανταγωνιστές μας που δεν υπάγονται στις ίδιες ε, πληροφορίες και όπως είπαμε, ακούσαμε και προηγουμένως, είναι πληροφορίες που ε, θεωρούνται εμπιστευτικές. Α, θα συμμορφωθείτε, λέει ο πρόεδρος, πάντως, με, αν αλλάξει νομοθεσία. Ωραία. Ε, ο εισηγητής, ε, προς την οικία είχατε μία ερώτηση. Ναι, θέλω μόνο να μου επιβεβαιώσετε αν η θηγατρική και η ΣΑΣ έχει κάνει φορολογική συμφωνία με τις φορολογικές αρχές του Λουξεμβούργου, χάρη στο οποίο έγινε ομιλική χρηματοδότηση ε, ρίχνοντας το στελεστή από το 29,4% στο 2,3% και στο Λουξεμβούργο. Πώς γίνεται αυτή η εσωτερική χρηματοδότηση, πόσους έχετε, πόσους υπαλλήλους έχετε στη θηγατρικές σας στο Λουξεμβούργο ε, και για την ε, δημοσίευση των εκθέσεων αναχώρα είναι πολύ σημαντικέ πληροφορίες για να ξέρουμε ότι καταβάλλεται ο φόρος εκεί που δημιουργείται η προσθέμενη αξία, εκεί που υπάρχει παραγωγή. Μπορείτε να το σχολιάσετε. Ευχαριστώ. Απάντηση. Interfinances, ε, ε, η ενδομιλική χρηματοδότηση. Αυτό είναι τμήμα των εσωτερικών διεργασιών ε, χρηματοδότησης μαζί και με την ελβετική θηγατρική Ευτυχώς έχουμε μετρητά. Με αυτή τη ρευστότητα και ε, βλέποντας ε, τι έγινε με την χρηματοπιστωτική κρίση, διαπιστώσαμε ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη ρευστότητα που έχουμε για να επεκταθούμε διαφορετικό τρόπο. Λοιπόν, διαχείριση των μετρητών και εσωτερική χρηματοδότηση αυτό είναι απαραίτητο για μια εταιρεία που έχει διασυνοριακές επιχειρήσεις. Τώρα, το, η δομή, μηχανισμός που έχουμε για τις, ε, την ενδομηλική χρηματοδότηση ε, απασχολεί συνολικά 10 ανθρώπους. Κάποιοι είναι στο Λουξεμβούργο και στην Ελβετία. Αληθεύει ότι επ' αυτών των ροών χρημάτων, όπως το υποδείξατε κι εσείς, είναι χαμηλή η φορολόγηση. Όλα τα αυτά είναι τέτοια οικονομική πραγματικότητα ε, που σε, αυτές τις, ε, σε αυτά τα τμήματα δεν έχουμε υψηλά κέρδη. Ε, μπορώ και να σας πω συγκεκριμένα περί πρόκειται. 10-15 εκατομμύρια το χρόνο. Αυτά εξοικονομούμε από το περιθώριο. Αλλιώς θα τα είχαμε δώσει σε ε, council, σε εταιρείε συμβούλων ε, για χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Αυτά κερδίσαμε μόνο, εξοικονόμησαμε. Ευχαριστώ. Ο Γκούναρ Χιόκμαρκ ε, για το ΕΛΚ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είμαι και πελάτη σας, λέει ο Πρόεδρος. Ναι. Θέλω να κάνω μια ερώτηση στο ΙΚΕΑ. Σε ΙΚΕΑ, ορίστε. Θα μπορούσα ε, να πω και στο McDonald's γιατί έχουν ισχυρή παρουσία στη Σουηδία, αλλά θέλω να ρωτήσω κάτι την IKEA. Μα κάνει εντύπωση ότι συνήθω εδώ στο Κοινοβούλιο, σε τέτοιε επιτροπέ. Ε, καλούμε κόσμο να έρθει να ε, κάνει, να καταθέσει μαρτυρία του και του ε, ασκούμε κριτική επειδή δεν ακολουθούν του κανόνε. και τώρα του ασκούμε κριτική και τους ε, καταδιώκουμε επειδή τηρούν του κανόνε και είμαστε και νομοθέτες. Ερχόμαστε δηλαδή και κατηγορούμε εταιρείε επειδή είναι νομοταγεί. Ε, για νόμους που εμείς με τον ΑΒ τρόπο έχουμε ψηφίσει. Και ήθελα να ρωτήσω την ΙΚΕΑ. Πώς πιστεύετε ότι η Ευρωπαϊκή Φορολογική Νομοθεσία επηρεάζει τις δραστηριότητε και την ανάπτυξη της εταιρείας IKEA που είναι από τις πιο... Ε, επιτυχημένες. Είναι ενδιαφέρον αυτό. Επίσης, πώς βλέπετε τις διαφορές ανάμεσα ε, στη γενική φορολόγηση σε άλλες περιφέρειες του κόσμου, σε σύγκριση με την Ευρώπη. Λατινική Αμερική, Ηνωμένε Πολιτείε, Ασία, Αφρική, γιατί είστε παγκόσμια εταιρεία, πολυεθνική. Και τέλος, πώς ε, βλέπετε τις συνέπειες των όσων πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την καταπολέμηση του BEPS. Δηλαδή, ε ε, λέει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα προχωρήσει περαιτέρω από άλλες περιοχές του κόσμου στην Ευρώπη. Πώς τα βλέπετε όλα αυτά, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Ελπίζω σωστά να το σημείωσα. Τέσσερις ερωτήσεις κάνατε. Για μένα είναι σημαντικό να πω ότι εκπροσωπώ την Inter IKEA που είναι εκείνος που είναι της ε, franchises ε, για την IKEA. Έχουμε συμφωνίες με πολλές εταιρείες ε, παγκοσμίω που δραστηριοποιούνται τοπικά. Ξέρω τι γίνεται στην Ευρώπη, αλλά στην Κίνα, στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι περιορισμένες οι γνώσεις μου. Θα έλεγα όμως ότι μπορούμε ε, να πούμε το εξής. Όταν παίρνουμε μια απόφαση βασιζόμαστε στην ε, καλή επιχειρηματική ε, απόφαση. Συνυπολογίζουμε και τους φόρους βεβαίως όταν παίρνουμε μια απόφαση επιχειρηματική, αλλά ποτέ δεν είναι ο κύριος λόγος για να λάβουμε μια απόφαση τα φορολογικά ζητήματα. Ε, στη συνέχεια, σε ό,τι αφορά τη φορολογική νομοθεσία και αυτά που προτείνονται ως κατευθύνες γραμμές των ΩΣΑ και τα ΜΠΕΠΣ, που είναι η διάβρωση ε, της βάσης και η μετατόπιση των κερδών, θα πρέπει πρώτα να δούμε ε, όλες τις προτάσεις παντού και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μην έχουμε επιπλέον περιπλοκές. Βεβαίως οι λύσεις δεν θα πρέπει να δημιουργούν περισσότερη γραφειοκρατία από όσοι χρειάζεται. Και τρίτον, είναι σημαντικό όταν έχουμε διενέξεις να υπάρχει ένας μηχανισμός που να μπορεί να τις διαχειρίζεται και να επιλύει διαφορές ε, μεταξύ διαφόρων κρατών για τη φορολογία. Δεν ξέρω αν απάντησα σε ερωτήσεις σας. Μήπως να επανέλθετε για τα ευρωπαϊκά ζητήματα. Ναι, αν, δούμε τι κάνουμε εμείς που είναι να δίδουμε το franchising, η βάση είναι στις κάτω χώρες, εδώ και 30 χρόνια και πλέον είναι βασική ε, δραστηριότητα με κάποιους εργαζομένους και μπορείτε να καταλάβετε ότι είναι σημαντικό αυτό. Δεν χρηματοδοτούμε, πώς να το πω, δεν επενδύουμε σε κτίρια και τα λοιπά, σε υποδομές, λόγω ε, κάποιης προλογικής νομοθεσίας. Δεν είναι αυτό το κίνητρο. Ευχαριστώ. Από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες, ο κύριος Εμμανουέλ Μογέλ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, σε ποιον απευθύνεται την ερώτησή σας, στη McDonald's. McDonald's γιατί είναι εξαιρετικό που έχουμε δυνατότητα να ξαναδούμε την εκπρόσωπο της McDonald's ε, κύριε Πρόεδρε. Είχα την δυνατότητα πριν από μερικές εβδομάδες ε, να υποβάλω ερωτήματα στη McDonald's και θέλω τώρα να αποσαφηνήσουμε κάποια πράγματα. Ε, μιλάμε για profit sharing υπέρ των εργαζομένων. όταν σας είχα κάνει την ίδια ερώτηση την προηγούμενη φορά μας είπατε ότι δεν καταλαβαίνετε ακριβώς περί τίνος πρόκειται. Είδαμε όμως ξαναείδα τα στοιχεία 20 ε, εκατομμύρια ε, μοιράζονται οι έξι επικεφαλής διευθυντές. Απ' την άλλη πλευρά ε, βλέπετε, λέτε ότι οι δυνατότητες που σας δίνουν τα δικά σας εστιατόρια είναι αυτά τα οποία δίνουν τη δυνατότητα για τέτοιους μισθούς κτλ. Όμως, όμως τα κέρδη των εστιατορίων περνούν μέσω... Έχετε δημιουργήσει μια εταιρεία πνευματικής ιδιοκτησίας η οποία δίνει τα Ρόγελτης στο Λουξεμβούργο και ε, μετά ε, επανέρχονται στην Ευρώπη μέσω της Ελβετίας. Επανέρχομαι λοιπόν πώς αυτές ε, οι, πώς αυτές οι θυγατρικές γίνονται ελληματικές. Ποια είναι η διαδικασία βάση της οποίας γίνονται ελληματικές και επομένως δεν έχετε επιστροφή κερδών. Απάντηση. Thank you for the question. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση όσον αφορά το profit sharing, ε, το σύστημα που εφαρμόζουμε στην McDonald's, εμείς πιστεύουμε ότι το σύστημα franchising που έχει η McDonald's δίνει ισχυρά ε, κίνητρα και κέρδη στην, ε, στους franchisees και επιτρέπει έναν ικανοποιητικό καταμερισμό ε, ε, κερδών. Από την άλλη πλευρά, όταν είναι κερδοφόρα μία επιχείρηση, ε, αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι έχουμε σε πέντε χρόνια δώσει 2,5 δις δολάρια σε corporate tax και επομένως θεωρώ ότι αυτό ήδη είναι ένα σαφές δείγμα. Όσον αφορά αυτό το ζήτημα για το Λουξεμβούργο. Αυτό που είναι σημαντικό να καταλάβει κανείς, ε, ε, μπορώ να σας δώσω βέβαια πληροφορίες για το Λουξεμβούργο, α, α, αλλά νομίζω ότι αλλού είναι το ζήτημα. Το Λουξεμβούργο ε, είναι έδρα ε, της εταιρείας η οποία δέχεται τα ρόγιαλ της, της πνευματικής ιδιοκτησίας του ονόματος κτλ οι franchisees έχουν την πρόσβαση ε, στο, ε, ε, στο brand name αλλά η McDonald's έχει και άλλα εισοδήματα από ιδιοκτησία ας πούμε και ακριβώς αυτό το σύστημα των franchisees μας δίνει το συγκριτικό πλεονέκτημα που μας επιτρέπει να έχουμε αυτό το κέρδος και βεβαίως εγώ δεν δέχομαι, δεν δέχομαι ε, με όλο το σεβασμό αυτό που λέτε όσον αφορά ε, την δημιουργία ελληματικών εταιριών κτλ. Κύριε Μορέλ, φοβούμε ότι, ε, φοβούμε ότι δεν, δεν καταλάβατε καλά. Ρωτώ λοιπόν, θεωρείτε ότι είναι λογικό ή οι διευθυντές σας να ε, έχουν τόσο μεγάλους μισθούς τη στιγμή που οι μισθωτοί σας ε, στις εταιρείες, στις θηγατρικές σας ε, που είναι αυτοί οι οποίοι σας φέρνουν τα χρήματα ε, δεν, δεν έχουν αντίστοιχα, ε, ε, αντίστοιχο επιμερισμό των κερδών. Αυτό σας ρωτάω. Γίνονται ελληματικές ή θυγατρικές σας έτσι ώστε να μην έχετε να δώσετε μετά τμήματα των κερδών στους franchisees. With respect to the salaries of... Όσον αφορά τους μισθούς ε, των ε, επικεφαλής μας, κοιτάξτε, αυτά αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, από το Board of Directors. Δεν έχω καμία ανάμειξη και δεν μπορώ να αναφερθώ σε αυτό. Όσον αφορά τώρα τις εργασιακές μας πρακτικές, ε, κοιτάξτε, πρέπει να σας πω ότι εμείς, εμείς έχουμε 420.000 απασχολούμενους ε, μέχρι των ε, συστημάτων ε, franchising και έχουμε, και έχουμε τη δυνατότητα να δημιουργούμε διαρκώς θέσεις εργασίας μέσω αυτών των, αυτών των εστιατορίων. Η McDonald's προσπαθεί ειλικρινά να είναι καλός εργοδότης. Πληρώνουμε ε, ε, ε, λογικούς μισθούς τα τελευταία χρόνια. Έχουμε βελτιώσει τις πρακτικές μας και τις πολιτικές μας. Επίσης έχουμε σταθερό feedback από τους ε, ε, εργαζόμενούς μας και προχωράμε σε διαφοροποιήσεις και προσαρμογές οποτεδήποτε παρουσιαστεί ανάγκη. Άρα υπάρχει, λέει ο Πρόεδρος, ένα διτό πρόβλημα. Το ένα είναι το εργασιακό, το άλλο είναι το φορολογικό. Ε, και ε, υπάρχει και το δεοντολογικό ερώτημα ε, των, της βελτιστοποίησης των φόρων και του κατά πόσον είναι δεοντολογικά σωστό αυτή η τόσο πολύ μεγάλη, αυτό το τόσο ψηλό μισολογικό καθεστώς για να το θέσω διπλωματικά. Από το ECR. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Μια ερώτηση για την οικία. Ο κώδικας ε, δεοντολογίας ε, της IKEA ε, είναι πολύ καλό ανάγνωσμα. Λέει στους εργαζόμενους ότι η IKEA είναι μια εταιρεία υψηλών ηθικών στάνταρ. Ρωτώ, είναι ηθικό, είναι νόμιμο το γεγονός ότι το ότι δουλεύετε για την IKEA ε, έχετε την δυνατότητα να ε, ε, σταθείτε απέναντι σε όσους ενδεχομένως κατηγορούν την IKEA έχετε την δυνατότητα να αποκαταστήσετε την αλήθεια όσον αφορά ε, τα τεχνάσματα τα φορολογικά γιατί σύμφωνα με μελέτες και με μια πρόσφατη έρευνα των πρασίνων ε, τα τελευταία έξι χρόνια πάνω από ένα δις ε, έχει ζημιωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι φορολογικές της υπηρεσίες ε, δεν πρέπει να αρχίσετε να πληρώνετε περισσότερους φόρους ε, εκεί που λειτουργείτε και έχετε έδρες. Δεν πρέπει να, δείξετε έμπρακτα την ε, στήριξή σας και την υποστήριξη των ηθικών αρχών μέσω προσαρμογής της συμπεριφοράς σας. Κύριε Διευθύνοντα Σύμβουλα, έχετε το λόγο. αν θέλουμε να αναλάβουμε ε, δημόσια την ευθύνη μας. Μα η παρουσία μου εδώ απαντάει ε, στο ερώτημά σας. 15 μισό πληρώνουμε σε φορολογικό συντελεστή για τους, ε, στους ενοποιημένους λογαριασμούς. Έχουμε κώδικα δεοντολογίας για τους ε, συνεργάτες μας, για τους ε, προμηθευτές μας, για τους καταναλωτές μας. Και φυσικά εξακολουθούμε να βελτιωνόμαστε. Και ε, δεν πρόκειται να τελειώσει, δεν έχει πέρασει αυτή η διαδικασία. Συνεχίζεται, σαν Υπάρχει και αυτή η έκθεση Είπατε υποτιθέμενη ε, η έκθεση. Είπα so-called green, υποτιθέμενη πράσινη έκθεση. Ε, ο κύριος, ε, κύριε Λάμπερς δεν έχετε το λόγο, θα τον πάρετε μετά. Ναι, τη διάβασα την έκθεση λοιπόν. Και μπορώ να σας δώσω και δύο παραδείγματα αβάσιμων ισχυρισμών και στην ε, περίληψη και στα εισφαλμένα ως εκ τούτου συμπεράσματα ότι πληρώνουμε τέλος franchising σε εμά τους ίδιους, αναφέρει η έκθεση. Δεν ευσταθεί αυτό. Έχουμε 13 ομίλους με franchisees που ε, ε, πληρώνουν τέλος in systems VV στην κεντρική εταιρεία όχι στους άλλους που έχουν επίσης franchise δηλαδή. Από το 83 δεν έχουμε franchise στην Ολλανδία και ε, διαπιστώσαμε ότι για την ε, άνθηση της επιχείρησής μας της ε, φιλοσοφίας IKEA και της ενίσχυσης παρουσίας μας παγκόσμιας, αυτός ήταν ο καλύτερος τρόπος με το franchising. Δεύτερον, μέσα στην ε, περίληψη της έκθεσης αναφέρεται το εξής, ότι χρησιμοποιούμε ένα ε, κανάλι πληρωμών, conduit λέει για τις ε, πληρωμές, αλλά φαίνεται ότι είναι μια οντότητα διέλευσης. Και κάποια πράγματα δεν συμβάλλουν ε, στην ανάπτυξη της IKEA και στην ενίσχυση της παγκόσμιας παρουσίας του. Ε, το IKEA Systems VV λοιπόν έχει πολύ συγκεκριμένε ε, και σημαντικέ δραστηριότητε στην Ολλανδία, κατάρτιση προσωπικό κτλ. Και το προσωπικό είναι πάνω από χίλια άτομα και κάνουν αυτή ακριβώ τη δουλειά. Ευχαριστούμε. Φάμπιο Ντεμάση για την γκουα θα πάω να κάνω barbecue με burger, με burgers, δηλαδή θα μιλήσω για το McDonald's γιατί ο φίλος μου ο Λάμπερς ειδικεύεται στην IKEA. Ε, σας ρωτήσαμε σε την προηγούμενη φορά για την παρουσίαση στους φορολογικούς παραδείσους και είπατε ότι μόνο για να πουλήσουμε χάμπουργκες θα ήμασταν σε αυτές τις χώρες. Και όταν μιλάμε για τις οντότητες και τους φορολογικούς ε, παραδείσους, ξεχάσατε να αναφέρετε τις Βερμούδες. Φαίνεται όμως ότι έχετε πολλές θηγατρικές και χάμπουργκερ δεν υπάρχουν εκεί, δεν πολλούνται, δεν έχετε ε, υποκαταστήματα γιατί είναι παράνομο παρά μόνο στην Αμερικανική στρατιωτική βάση της Βερμούδας ήταν αυτό δυνατό, αλλά έκλεισε η βάση το 1995. Γιατί παραλείψατε το, τις Βερμούδες και τι κάνετε εκεί, εν πάση περιπτώσει, αν δεν πουλάτε μπέργκερς. Αφήστε που δεν μιλήσατε για τη φορολογική συμφωνία με το Λουξεμβούργο. Μιλάτε για τα chicken nuggets, τα κομματάκια κοτόπουλο, μιλάτε για τα χάμπουργερ, αλλά για τη φορολογική συμφωνία κουβέντα. Έχω άλλα 45 δευτερόλεπτα. Ε, Ελβετία και Delaware. Έχετε στο Λουξεμβούργο το μεγαλύτερο franchising ε, για την Ευρώπη. Και ε, πριν πάνε στη ΣΥΠΑ τα κεφάλαια περνάνε μέσα από την Ελβετία. Γιατί γιατί περνάνε από την Ελβετία και μετά επιστρέφουν στην Delaware, στη ΗΠΑ. Για σας πω γιατί, διότι ε, ισχύει εκεί εξαίρεση για τα φορολογικά έσοδα και είναι μηδενικό ο συντελεστή στην Ελβετία. Γι' αυτό έχετε αυτή την περίπλοκη ρύθμιση. Και πρέπει να πάρω τον Μπέρνι Sanders για να μπορέσει να αλλάξει κάτι επιτέλους αυτή την κατάσταση. Ευχαριστώ. Το Νοέμβρη δεν είχαμε καμία διάθεση να παραπληροφορήσουμε την, Ευρω... την Επιτροπή. Σωστά είπαμε ότι έχουμε 230 εστιατόρια και 10.000 αποσχολούμενους στην Ευρώπη. Οι υπόλοιποι είναι franchises, είναι ανεξάρτητοι σε πολύ περιορισμένο ρυθμό περιπτώσεων έχουμε, ε, έχουν κάποιοι franchises και ε, ακίνητα τα οποία όμως δεν έχουμε στην ιδιοκτησία μας τα χρησιμοποιούν για τα εστιατόρια, για τις βερμούδες παρότι το McDonald's είναι μέσα ε, στο όνομα, στην εταιρική επωνυμία δεν διοικείται από τις ΙΠΑ. Διακόπτει ο κύριος Ντεμαζή. Τι κάνετε εκεί πέρα, ασφαλίζετε χάμπουργκες, ε, τι κάνετε ακριβώς. Απάντηση. Μα είναι ήδη ασφάλισης και αντασφάλισης δεν μπορώ να σας δώσω τις λεπτομέρειες τώρα αλλά μπορώ συγκεκριμένα γραπτός να σας στείλω τις ε, λεπτομέρειες για αυτά που κάνουμε στις ε, Βερμούδες κανένα πρόβλημα, θα τα, στείλω στην Επιτροπή και θα τα διαβιβάσουν. Την Ελβετία, δεν μου απαντήσατε για την Ελβετία. Λοιπόν, να τον κόσμο οι πολιεθνικές ανάλογα με τις δραστηριότητες, ανάλογα με τα νομικά συστήματα και άλλες παραμέτρους σχεδιάζουμε τους μηχανισμούς μας ώστε να λειτουργήσουμε σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Το McDonald's διαπίστωσε ότι ε, πρέπει να αναδιαμορφώσει την εταιρική του δομή ώστε να ταιριάζει με το επιχειρηματικό μας μοντέλο για κάποιες συγκεκριμένες περιοχές. την Ελβετία τη επιλέξαμε, διότι εκεί μπορούμε να συγκεντρώσουμε κάποιους από τους βασικούς ηθήνοντες. Διακόπτω κύριο Ντεμάζη. Μου θυμίζετε την εξάχρονη κόρη μου όταν πρέπει να πει το ποίημα, ε, γιο όταν πρέπει να πει το ποίημα για το νηπιαγωγείο. Ε, δεν θέλω να μου απαγγείλετε, θέλω να μου πείτε τι κάνετε στην Ελβετία. Δεν γιατί πάνε τα χρήματα στην Delaware μετά την ε, Ελβετία. Ναι, η δομή ο μηχανισμός στο Λουξεμβούργο έχει υποκατάστημα στην Ελβετία, αλλά αυτό είναι ε, υποκατάστημα της εταιρείας ε, της Αμερικανικής. και είπαμε ότι υπάρχουν ε, διαφορές στα συστήματα. Έχουμε κατευθυντήριες γραμμές ε, για την καινοτομία στρατηγική. Δεν έχει καμία σχέση με το Ρόγελ αυτό που έχουμε στην Ελβετία. Δηλαδή η Ελβετία δεν παίρνει τα Ρόγελ Υπάρχει διοικητική λειτουργία αλλά δεν έχει καμία σχέση η Ελβετία με τα royalties. Ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος, και γι' αυτό το σημείο θα θέλαμε να μας στείλετε γραπτός. Ναι, ναι, λέει ο κ. να πάρω τηλέφωνο τον Μπέρνι Σάντες. Θα εξετάσουμε το αίτημά σας. Γιατί είναι περίπλοκο, λέει ο πρόεδρος, και δεν έχουμε και, και χρόνο. Χρειαζόμαστε πάντως λεπτομέρειες. Είναι σημαντικό για τα μέλη της Επιτροπής μας. Και τώρα θα δώσω το λόγο στον υποτιθέμενο πράσινο Φιλίπ Λαμπέρτς και να απαντήσω και εγώ στον υποτιθέμενο πρόεδρο με χαρά και να κάνω μια ερώτηση στην υποτιθέμενο ε, εκπρόσωπο της υποτιθέμενης εταιρείας IKEA προηγουμένως. Κύριε Γιάννη και κύριε Χάνσε, σίγουρα σας νοιάζουν ε, οι δουλειές, οι θέσεις εργασίας και ιδιαίτερα η δικιά σας. Και θα ήθελα να σας προειδοποιήσω ότι η σημερινή σας επίδοση ε, γενικά στη συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη ε, δίνει ε, περισσότερη ε, αξιοπιστία στο επιχείρημα ότι ακριβοπληρωμένες θέσεις όπως οι δικές σας μπορούν να αντικαταστηθούν από κομπιούτερ. Διαβάζετε σαν μηχανές κείμενα που έχετε που θα μπορούσε να διαβάζει ένα ρομπότ ή ένα κομπιούτερ. Εσείς αυτά τα ακούτε που λέτε, τα συνειδητοποιείτε, προσοχή, γιατί μπορεί να σας βγει μπούμεραγκ. Κύριε Χάνσεντ, λέτε ότι πληρώνετε 15,5% φορολογικό συντελεστή για το Inter-IKEA Group, τον όμιλό σας, για να καταλάβω δηλαδή. Η εταιρεία σας 3% ε, του τζίρου, όχι ε, των ε, κερδών, παίρνει από όλους τους franchisees. Στην Ολλανδία πηγαίνουν τα λεφτά αυτά σε κάτω χώρες και μετά ένα σημαντικό κλάσμα στο Λουξεμβούργο, το 1 τρίτο, και δεν είναι και πολλά τα λεφτά, σε αγνώστους δικαιούχους. Πού είναι το 15% στο υπόλοιπο, φορολογείται το σύνολο, αφού έχετε διαβρώσει τη βάση σε μεγάλο βαθμό και κατά τα άλλα θα πρέπει να συνεργάζεστε καλά με την Interco Finance γιατί έχετε τον ίδιο οικονομικό διευθυντή. Τουλάχιστον οι δύο ε, θα πρέπει να συμφωνούν. Ε, ε, στο Λουξεμβούργο λοιπόν, τα λεφτά που πάνε εκεί ε, είναι, πληρώνουν φόρους, ε, συγγνώμη, τόκους. Ε, ξέρετε αυτό, έχετε και ένα ruling με το Λουξεμβούργο και πληρώνετε 0,0 κάτι της εκατό που είναι σχεδόν ε, κοντά στο μηδέν. Εγώ είμαι μηχανικός και ξέρετε τα στρογγυλεύω τα ποσά. και τα λεφτά πάνε στο Λίχτενστάιν μετά, που είναι μια ωραία χώρα, πλην όμως δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επειδή είμαι και χαζός και δεν μπορεί να με αντικαταστήσει μηχανή, γιατί τα μηχανήματα είναι τουλάχιστον ε, νοήμονα, έστω και τεχνητή νοημοσύνη. Ολλανδία, Λουξεμβούργο, Λίχτενστάιν Τι το ιδιαίτερο έχουν αυτές οι χώρες για να πάτε εκεί, αν όχι πολύ ε, ευνοϊκές φορολογικές ρυθμίσεις στην νομοθεσία. Και ένα τελευταίο, όταν λέτε, δεν θυμάμαι ποιος το είπε από τους δυο σας, ότι οι νομοθέτες νομοθετούν και εμείς συμμορφωνόμαστε και υλοποιούμε. Επιτρέψτε μου να διαφωνήσω λίγο και εσείς και η Business Europe, αν δείτε πόση ενέργεια βάζετε για να επηρεάσετε την νομοθετική διαδικασία σε διάφορες χώρες στην Ευρώπη, θα έλεγα ότι τουλάχιστον έχετε βάλει και εσείς το χεράκι σας στους, για να γίνουν αυτοί οι, δρόμοι, οι νόμοι που ισχυρίζετε στη συνέχεια ότι ε, υλοποιείται. Και δεν θέλω να μου τα πείτε σαν μηχανήματα, σαν πραγματικοί άνθρωποι θα σας ήμουν ευγνώμη και θα ήταν ωραίο. Ένα λεπτό και 20 τώρα έχουν οι άνθρωποι για να απαντήσουν. Οικαία οι λάθος παραδοχές οδηγούν και σε, εσφαλμένες, ε, σε εσφαλμένα συμπεράσματα καμιά φορά. Το 3% του τζίρου που πληρώνουν όλοι όσοι έχουν το franchise ως τέλος δεν είναι ε, αφαίρεση κερδών σε όλες τις franchise παντού στον κόσμο έχουν τη δυνατότητα και το δικαίωμα να πολλούν IKEA σε καταστήματα IKEA να χρησιμοποιούν τη φύρμα ε, και υπό την ε, ε, συνολική φιλοσοφία της IKEA. Κάνουν business και δραστηριοποιούνται και πληρώνουν πολλούς φόρους στις χώρες τους. Η Inter IKEA που εκχωρεί το franchise δρεύει στις κάτω χώρες από το 1983 και είναι ο τελικός αποδέκτης του τέλους αυτού για να χρησιμοποιείται το εμπορικό σήμα ο όμιλος Interigea που εγώ εκπροσωπώ, Interigea Group, 15,5% πληρώνει ε, σε ε, ενοποιημένους φόρους. Κάνατε μια ερώτηση για ε, την εταιρεία στο Λουξεμβούργο. Και εμείς είμαστε σε μια διαδικασία διευκρίνησης και απλούστευσης. Το 2012 Ε, αγοράστηκαν για 9 δις ευρώ ε, δικαιώματα πνευματικά που έχουν να κάνουν με το εμπορικό σήμα. Και ο ιδιοκτήτης μας και το Ίδρυμα στο Λίχτενστάιν ε, έδωσε πολύ κεφάλαιο, 3,6 δις ευρώ και το υπόλοιπο δόθηκε από τον ιδιοκτήτη μας μέσω ενός δανείου όπου προφανώς θα πρέπει να πληρώνουμε τόκους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την ε, υποτιθέμενη απάντηση. Ε, αυτό που προτείνω να γίνει τώρα εδώ, γιατί υπήρξε και έκθεση πάρα πολύ εμπεριστατωμένη και πάρα πολύ συγκεκριμένη και ακριβής που κατατέθηκε υπό την πολιτική ε, ηγεσία και πρωτοβουλία των Πρασίνων. Να απαντήσει γραπτός ε, όμιλος IKEA και να πει ε, τι, τα, ποια είναι τα σημεία με τα οποία συμφωνεί και ποια αμφισβητεί. Και δεν είναι καθόλου μηχανές, είναι άνθρωποι υπεύθυνοι και ο καθένας φέρει την ευθύνη του αγαπητέ συνάδελφοι. Λοιπόν, θα δώσω τώρα το λόγο στο Μάρκο Τζάνι, εξ ονόματος της ομάδας. Ευχαριστώ. Στον εκπρόσωπο της IKEA θα ε, ρωτήσω κάτι. Θα ήθελα ε, και εγώ, όπως και οι συνάδελφοι που μίλησαν προηγουμένως, να επικεντρωθώ σε ένα σημείο. Έχω την εντύπωση ότι δεν υπάρχει αρκετή σαφήνεια ή τουλάχιστον ε, οι απαντήσεις, ακόμα και η τελευταία που μόλις ακούσαμε, δεν με ικανοποιούν. Όσον αφορά την δομή σας στο Λουξεμβούργο, τα στοιχεία LuxLeaks είναι σαφή εγώ θέλω να μιλάω με αριθμούς ε, και στην ίδια την έκθεση της Price Water ε, η οποία Price Water Cooper ε, η οποία είχε υπογράψει το χαρτί αναφέρει ότι 48.000 ευρώ ε, πληρώθηκαν ε, σε, για φόρους ε, για, για κέρδη πάνω από 2 δις. Είναι κάτω από το 1%. Είναι 0,0 κάτι το ποσοστό. Ε, και σας ρωτώ, αυτά, αυτά τα στοιχεία, λαμβάνοντας υπόψη ότι προέρχονται από συγκεκριμένα επίσημα χαρτιά της White House ε, Cooper, είναι ε, και που ήταν ο φοροτεχνικός σας σύμβουλος. Αυτά τα στοιχεία λέω τα επιβεβαιώνετε. Ένα άλλο στοιχείο το οποίο ε, προέρχεται πάλι από τα ίδια στοιχεία και που αφορά αυτήν την ε, ταμιακή σας δομή στην Ευρώπη μέσα από υβριδικές μορφές ε, που επιτρέπουν την μη διπλή ε, φορολόγηση των ενδοομιλικών δανείων έχουν οδηγήσει ε, σε ε, πληρωμή 2 εκατομμυρίων σε φόρους για αυτά τα δάνεια εντός του ομίλου ε, για δάνεια 35 δις. Επομένως θα θέλαμε, αυτά είναι στοιχεία τα οποία η φοροτεχνική σας, οι σύμβουλοι σας έχουν επιβεβαιώσει και γνωστοποιήθηκαν μέσω των διαρροών LuxLeaks. Απάντηση. Εγώ εκπροσωπώ τον όμιλο Ιντερικέα. Ρωτήσατε δύο πράγματα. Το ένα που σχετίζεται ε, ε, σχετίζεται με τον ιδιοκτήτη και ένα που σχετίζεται με, την, με τον όμιλο Ιντερικέα. Όσον αφορά τα tax rulings ε, του Λουξεμβούργου από το 2001, όπως είπατε προηγουμένως, όντως υπήρξαν κάποιες αποκαλύψεις. Το ruling του 2009 αφορά, σχετίζεται με κάποιες αλλαγές στον νόμο του Λουξεμβούργου και κάποιες δικές μας αλλαγές. Στόχος του ruling αυτού ήταν να ε, ήταν ε, να επιβεβαιώσουμε την ορθή από τη δική μας πλευρά ερμηνεία των πραγμάτων. Ε, εμείς πάντα συμμορφωνόμαστε με τους κανονισμούς και με τους νόμους οπουδήποτε είμαστε παρόντες. Η Finance SA Luxembourg όντως, όντως έχει πληρώσει φόρο της τάξεως ποσοστό δηλαδή φορολογίας τάξεως 2%. Δεν είναι σωστά τα αριθμητικά στοιχεία τα οποία δώσατε. Το συνολικό ποσοστό όμως του ενοποιημένου φόρου ε, για το Inter Ikea Group ξεκινάει από το 14% και φτάνει μέχρι το 17%. επιπλέον των φόρων που πληρώνουμε σε αυτά τα πλαίσια πληρώνουμε και άλλους ε, φόρους που αφορούν την κερδοφορία ή ε, άλλα στοιχεία της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας. Όσον αφορά την υβριδική, ας πούμε, τα υβριδικά ε, μοντέλα, νομίζω ότι εδώ θα πρέπει να μου πείτε τι εννοείται υβριδικά μοντέλα φορολόγησης. Σε γενικές γραμμές αναφέρομαι σε intercompany κάνει δάνεια λαμβάνοντας υπόψη την ειδική μορφή, ε, ε, την ειδική ταμιακή μορφή που έχετε. Ε, ναι, κοιτάξτε, ο δανεισμός ε, ένθεν και ένθεν των ε, ε, διαφόρων πλευρών ας πούμε ενός ομίλου είναι μια συνηθισμένη διαδικασία. Έχουμε και μια διαχείριση ρευστού, cash management, το οποίο ακολουθεί συγκεκριμένους κανόνες. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να πληρώσουμε, να δώσουμε περισσότερα περιθώρια κέρδους σε άλλους, σε εξωτερικούς ή τρίτους παράγοντες ναι, είναι γεγονός ότι προσπαθούμε στα πλαίσια της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας να ε, διατηρήσουμε τα ποσοστά μας. Άλλη ερώτηση. Το ruling το οποίο διαπραγματευτήκατε με το Λουξεμβούργο του 2009 ε, βρίσκεται ακόμα σε ισχύ. ήταν θέμα ερμηνείας ε, του, του νόμου. Δεν ρωτάω αυτό, ρωτάω αν ισχύει ακόμα. Ναι, ισχύει ακόμα. Ο κύριος Άνεμανς από την ΕΝΕΦ. E Ευχαριστώ πρόεδρε. Ε, στα Ολλανδικά θα μιλήσω. Και προς τους δύο θέλω να ρωτήσω. Να το πάρω αλλιώ. Γιατί η σημερινή ακρόαση με όλες αυτές τις πολυεθνικές είναι το ίδιο τροπάρι. Ε, ε θεωρείτε ότι έχετε ηθική ευθύνη ή όχι, αλλά δεν μας λέτε πολλά περισσότερα από αυτά ότι πληρώνετε φόρους, ότι είστε πρόθυμοι, ότι έχετε μεγάλο ενδιαφέρον, έρχεστε εδώ για προθυμία και ε, ε, ε, διάλογο. Τα ακούμε από την αρχή της ακρόασης. Να το πάρω αλλιώ λοιπόν για να ρωτήσω το εξή. Με τον ΑΒ τρόπο προτιμάτε να διατηρηθεί το σημερινό σύστημα ή θέλετε να αλλάξει. Υπάρχει δυνατότητα για ένα άλλο σύστημα που θα σας βολεύει καλύτερα με βάση το επιχειρηματικό σας μοντέλο. Και αν ναι, ποιο είναι αυτό. Και δεύτερη ερώτηση, περιμένετε αλλαγές μετά το σκάνδαλο LuxLeaks, ε, τον τρόπο με τον οποίο τα θεσμικά όργανα τώρα ασχολούνται με αυτό το θέμα. Και έχετε ήδη προετοιμαστεί για τέτοιες εξέλιξεις. Okay. Madame. Ε, ε, κύριε Πτωμακτολάντς, ε, ναι. Σε ό,τι αφορά ε, τις μεταρρυθμίσεις σε σχέση με το σημερινό σύστημα, εμείς θέλουμε νόμους που να προάγουν τον ανταγωνισμό, αλλά να έχουν κάποια συνάφεια, κάποια συνέπεια, κάποια σταθερότητα και να είναι απλοί. Χαιρόμαστε πολύ και εκτιμούμε τις προσπάθειές σας, αλλά δεν κάναμε συγκεκριμένες προτάσεις. Περιμένουμε οι νομοθέτες να νομοθετούν και οι εταιρείε ε, να ε, συμμορφώνονται. Αυτό κάνουμε. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Άνσεν. As, as I mentioned... Όπως σας είπα προηγουμένως, ε, χαιρόμαστε πάρα πολύ και θα καλωσορίζαμε οποιαδήποτε πρωτοβουλία σχετικά που θα οδηγούσε σε απλούστευση μεγαλύτερη σαφήνεια για τις εταιρείες. Τώρα, θα πρέπει οι λύσεις να μην είναι πάρα πολύ βιογραφι... Ε, ε, γραφειοκρατικές και βαριές. Ε, δεν θέλουμε ιδιαίτερη επιβάρυνση. ξέρουμε ότι μια στοιχειότητα θα υπάρχει και είμαστε έτοιμοι να το αντιμετωπίσουμε. Από κοινού όμως επιχειρήσεις και νομοθέτες μπορούμε να κρατήσουμε τα πράγματα έτσι σε ένα απλό επίπεδο και αν το καταφέρουμε αυτό θα μας βοηθήσει όλους. Μάλιστα λέει ο Πρόεδρος. Σοσιαλιστές και Δημοκράτες, ο Σέρτζο Κοφεράτη παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ήθελα να ρωτήσω την ε, ε, ευγενιστάτη κυρία Γκιαίτσα. Εάν θυμάται τι έλεγε, τι έλεγε ο Ράι Κρόκ, ιδρυτής ε, της ε, McDonald's. Εμείς έχουμε υποχρέωση να επιστρέψουμε κάτι στις κοινότητες που μας δίνουν τόσα. Αναρωτιέμαι αν θα συμμεριζόταν την τωρινή φορολογική σας πολιτική, γιατί δεν φαίνεται να κάνετε πολύ μεγάλη επιστροφή. Ας μην μιλήσω δε για τις ε, συγκεκριμένες εργασιακές ε, πολιτικές ε, των εργαζομένων σας, αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα, δεν αφορά τη δική μας Επιτροπή. Στην τελευταία φορά που μιλήσατε ενώπιον της Επιτροπής μας, δεν είχατε καθόλου αναφέρει τις δύο tax rulings με το Λουξεμβούργο. Είχατε δύο tax rulings σύμφωνα με τις προ σύμφωνα με τα στοιχεία της ε, Επιτροπής μας, ε, σας έδωσαν τη δυνατότητα να αποφύγετε φορολόγηση, καταβολή φόρων δηλαδή, στο Λουξεμβούργο και στις Ηνωμένε Πολιτείε. Αναρωτιέμαι και ρωτώ ε, εξακολουθείτε να χρησιμοποιείτε τα tax rulings γιατί θεωρείτε ότι σας δίνουν ασφάλεια δικαίου ή γιατί κερδίζετε χρήματα. Εγώ θεωρώ βεβαίως ότι αυτά είναι παράνομα εργαλεία, ωστόσο τα έχετε χρησιμοποιήσει. Το δεύτερο, το οποίο θα ήθελα να σας ρωτήσω, αφορά τις ε, επαναλαμβανόμενες δηλώσεις σας σχετικά με την σημασία που αποδίδεται στην κοινωνική ε, υποχρέωση ή ε, ευθύνη της επιχείρησής σας. Αυτή η εταιρική ευθύνη, ας πούμε, το 2014 ε, παρουσιάσατε μία έκθεση για την ε, καλή επιχειρηματικότητα. Ωστόσο, δεν υπάρχει κανένα κεφάλαιο στα πλαίσια του γενικότερου κεφαλαίου για τις σχέσεις με την κοινωνία, καμία αναφορά λέω, στους φόρους που πληρώνετε Τώρα, μία κοινωνική ευθύνη η οποία δεν σχετίζεται ούτε με την εργασιακή ε, δικαιοσύνη ούτε όμως ε, και με τους ε, φόρους είναι λίγο ελαφριά, επιτρέψτε μου την έκφραση. Σας ευχαριστώ. Απάντηση. Ευχαριστώ που μου δίνετε την δυνατότητα να απαντήσω. Ήταν πολλές οι ερωτήσεις, θα προσπαθήσω να τις απαντήσω. Όσον αφορά την υποχρέωση να επιστρέψουμε κάτι στην κοινότητα, ναι, πιστεύουμε ότι το κάνουμε. Έχουμε τους ε, franchisers, δίνουμε, ε, παρέχουμε θέσεις εργασίας, κατάρτιση στα πλαίσια των, ε, των εστιατορίων μας ε, επίσης πρέπει να σας πω ότι συνολικά η McDonald's έχει πληρώσει 2 δις ε, και έχουμε ε, σε φόρους και έχουμε ένα μέσο όρο συντελεστή φορολογικού της τάξης του 30-31%. Ε, επίσης επανεπενδύουμε ένα τρίτο των ε, κερδών μας ε, και πιο εξειδικευμένα πρέπει να σας πω ξανά στα τελευταία πέντε χρόνια ο μέσος όρος του φορολογικού μας συντελεστή ήταν στο 27%. Νομίζω ότι είναι πολύ ψηλότερος από αυτόν τον μεμονωμένο συντελεστή πολλών κρατών μελών, πολλών χωρών της Ευρώπης. Εμείς βοηθάμε επίσης ε, τους ε, franchisees ε, με το ισχυρό brand name και με, του παρέχουμε ευκολίες πρόσβασης στο brand name αλλά και σε άλλες ευκολίες που παρέχει η εταιρεία και με αυτόν τον τρόπο λειτουργούμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Merci. Ναι, εγώ όμω αναφερόμουν σε κάτι άλλο. Εγώ δεν αναφέρομαι στην φιλανθρωπία ή στην φιλεύσπλαχνη πολιτική, αλλά όταν κάποιος παράγει ε, ο κέρδος ε, ε, επιστρέφει με δύο ιστορικά αποδεκτούς και σημαντικούς τρόπους. Με τις ισότιμες ε, και σωστές εργασιακές συνθήκες και την ταυτόχρονη σωστή αμοιβή των εργαζομένων αφενός και με την πληρωμή των οφειλωμένων φόρων αφετέρου. Τα υπόλοιπα όλα είναι στη σφαίρα της φιλευσπλαχνίας και της φιλάνθρωπης πολιτικής ε, κοιτάξτε, ε, ε, εγώ δεν λέω να μην κάνετε φιλανθρωπίε, αλλά πρέπει κυρίως να μην είστε άδικοι απέναντι στους εργαζόμενους. Αυτό είναι πολιτική αξιολόγηση, αγαπητέ φίλε. Ε, θα, χαίρομαι για την ευκαιρία που έχω να διευκρινίσω. Υπάρχουν πολλά στοιχεία βεβαίως για την εταιρική ευθύνη και τα φορολογικά ε, του Μακδόλαντ. κινδυνεύω να ε, επαναληφθώ 27% 2,5 δις ε, νομίζω αυτό δείχνει έντονη κοινωνική ευθύνη 450.000 25.000 μάλλον εργαζομένους έχουμε στην Ευρώπη έχουν και κατάρτιση 40 ώρες το χρόνο και έτσι μπορούν να ε, έχουν και νέα προσόντα και να προχωρούν και την καριέρα τους. Ωραία, ευχαριστώ πολύ για αυτές τις σημαντικές διευκρινήσεις. Νίντερ Μάγερ. Ζητώ συγγνώμη που σας ξέχασα προηγουμένως. Ευχαριστώ. Έχω ερωτήσεις και προς τις δύο εταιρείε. Χαίρομαι που ήρθατε. Εγώ δεν θα είμαι τόσο ευχάριστος όσο συνάδελφοι να καταλάβετε ότι είμαστε πάρα πολύ απογοητευμένοι από την παρούσα κατάσταση που δημιουργήθηκε από τους συναδέλφους στα Εθνικά Κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις και η κατάσταση ε, την οποία εκμεταλλεύτηκαν ε, σπόδρα ορισμένες εταιρείες. Θα ήθελα να μάθω τα σχόλιά σας για τη συγκεκριμένη πρόταση που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δεν πιστεύω ότι δεν τα έχετε μελετήσει πάρα πολύ ε, εκτενώς. Τρία σχόλια με ενδιαφέρουν ε, από αυτά που άκουσα από την ΙΚΕΑ και θα ήθελα να μάθω και τις απόψεις σας γι' αυτό. Επίσης να δω τι γίνεται με αυτά που είπε η κυρία από τα McDonald's ότι ανησυχείτε μήπως αποκαλύψετε κάποια στοιχεία για το CBC, ε, μήπως εκθέσετε την εταιρεία σας. Για το CBCR, ε, το μητρό δηλαδή των καταχωρημένων εταιριών και σε ό,τι αφορά την πρώτη περίπτωση θέλω να ρωτήσω τι γίνεται με τη δυνατότητα να εισαχθεί η κοινή ενοποιημένη βάση για τη φορολόγηση των επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να καταλάβετε ότι αν υπάρξει κάτι τέτοιο δεν θα είναι πάρα πολύ εύκολο. Και στις 28 χώρες μέλη Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα ε, ε, από τη μια χώρα στην άλλη, αλλά θα απλουστεύσει ε, την ζωή των εταιριών. Πώς φαντάζεστε μια τέτοια ε, κατάσταση, ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Σε ό,τι αφορά ε, την, ε, τις εκθέσεις αναχώρα, είμαστε υπέρ της πρότασης του ΩΣΑ. Βεβαίως θα πρέπει να είναι ε, εμπιστευτικές οι πληροφορίες. Το κόστος, το benchmarks και οι πελάτες είναι κάποια στοιχεία εμπιστευτικά για μας. Ε, αν όλοι είναι υποχρεωμένοι να μοιράζονται ε, όλες τις προφορίες, καλώς. Σε άλλη περίπτωση δεν υπάρχει ισότητα στους κανόνες του παιχνιδιού. Και ε, ε, για το CCTV, συγγνώμη, για αυτό το συγκεκριμένο, ο Λούντεκ θέλει να ρωτήσει κάτι άλλο. Μα... Η έκθεση αναχώρα είναι Πολύ απλή, γιατί ε, τι σας προβληματίζει, τι σας ενοχλεί. Δεν ξέρω ε, αν μπορώ να σας δώσω ένα συγκεκριμένο στοιχείο, αλλά πρέπει να ε, δίνουν οι ανταγωνιστές τα ίδια στοιχεία, ιδιαίτερα σε μια συγκεκριμένη οικονομία, σαν συγκεκριμένο κλάδο με τους ανταγωνιστές. Έχω δει διαφορετικούς τρόπους. 750 εκατομμύρια είναι μια εταιρεία ας πούμε, που πληρώνει φόρους, αν δημοσιεύσουμε τώρα όλα τα στοιχεία αναχώρα, αυτό θα είναι κάτι που θα χρησιμοποιήσουν και θα εκμεταλλευτούν οι ανταγωνιστές. Ο κύριος Άνσεν. Ευχαριστώ. Όπως έλεγα, ε, πρόσδεκτες όλες οι πρωτοβουλίες που οδηγούν σε απλούστευση για τις έκθεσεις αναχώρα. Δεν ξέρω ακριβώ γιατί μιλάτε για αυτό το πίνακα. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες σε όλες τις φορολογικές δικαιοδοσίες εφόσον εμείς υποβάλλουμε τη δήλωση τη φορολογική. Και από κεντρικό επίπεδο θα μοιραστούμε τις πληροφορίες, θα τις κοινοποιήσουμε. Το πιο σημαντικό είναι να είναι σωστές οι πληροφορίες που έχουν οι φορολογικές αρχές για να ερμηνεύσουν σωστά την νομοθεσία και να έχουν σωστές πληροφορίε για το φορολογικό βάρος. Δεν είμαι σίγουρος ότι αυτή τη στιγμή το να δημοσιεύονται οι πληροφορίες θα βελτίωνε την κατάσταση. Είπατε στην αρχή ότι έχετε τρία σχόλια για τα, το αντιμπέψε. Ναι, ε, θέλω να πω ότι είναι σημαντικό να υπάρχει ευθυγράμμιση και αποχώρηση εκτός Ένωσης. Δεύτερον, να μην είναι υπερβολική η γραφειοκρατία, που, η επιπρόσθετη δηλαδή, που θα δημιουργηθεί. Και τρίτον, όταν υπάρχουν διαφορές, να υπάρχει μηχανισμός επίλυσης των διαφορών. Ταχαίως για να συνεχίζουμε τις δραστηριότητες μας. Ναι, ναι, αυτά μας είπατε και νωρίτερα, λέει ο Πρόεδρος. Λοιπόν, Ελκ Πάμπλο Θάλμπα, Ντενουέβο. Ξανά λοιπόν. Ευχαριστώ αγαπητέ Πρόεδρε. Θέλω να κάνω μια ερώτηση που έκανα και προηγουμένως. Με επικοδομητικό πνεύμα. Είναι γεγονό ότι πολλές από τις ειδήσει που μαθαίνουμε προκάλεσαν, πώς να το πω τώρα, αν μη τι άλλο, ε, μια ταραχή στην ευρωπαϊκή κοινωνία και ένα άλλο ε, σχετικά με τις πρακτικές ορισμών εταιριών που μερικές από αυτές είδαμε σήμερα. Και βεβαίως υπάρχει λόγος να έχουμε θορυβηθεί. Και το κοινοβούλιο μας ε, συνέστησε τη συγκεκριμένη επιτροπή μας και κάνουμε συστάσεις που προτείνουν κάποια βήματα για να έχουμε μια πιο στενή φορολογική ένωση και σήμερα συζητούμε κάποιες πρακτικές. Θέλω να μου αξιολογήσετε τα βήματα που έχουν γίνει μέχρι τώρα και αν προτείνετε και τίποτα επιπλέον σε σχέση με αυτό που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και πάλι σε επικοδομητικό πνεύμα θέλω να σας ζητήσω μια ανάλυση για το πόσες, ε, πόσους φόρους μάλλον πληρώνω σε κάθε χώρα οι εταιρείε σας για ΦΠΑ, ποιο είναι η φόροι που πληρώνετε για τους εργαζομένους σα. τι ποσοστό αναλυτικά έχετε τα στοιχεία να μας τα δώσετε αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Και προς τους δύο λοιπόν ε, ήταν αυτή η ερώτηση, μάλιστα. Παρακαλώ κυρία Γέιτ. Ευχαριστώ. Δεν έχω τα στοιχεία για το ΦΠΑ ούτε για το φόρο εισοδήματος είναι υψηλέ οι πωλήσει μα, φαντάζεστε ότι και ο ΦΠΑ θα είναι ανάλογο. Εξαρτάται από το μέσο συντελεστή. Το ίδιο ισχύει και για τι κοινωνικέ εισφορέ και για του φόρου που πληρώνουν οι εργαζόμενοι μα. Ε, Εμεί δραστηριοποιούμεθα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και πληρώνουμε φόρου εκεί που ε, έχουμε την επιχειρηματική μας δραστηριότητα. Ε, σε ό,τι αφορά τα περισσότερα βήματα και ιδέες σας ευχαριστούμε για τις προσπάθειές σας και εμείς θα καλωσορίσαμε οτιδήποτε ε, βοηθάει θα πρέπει να υπάρχει μια ενιαία πρόταση που να μειώνει την ε, περιπλοκότητα και να κάνει το σύστημα πιο συνεπές, πιο σταθερό και πιο σαφές και πιο απλό. Μπορώ να προσθέσω κάτι, λέει ο Πρόεδρος. Σε, κάτι, σε αυτό που ρώτησε ο Πάμπλο για τις συστάσεις που θα μπορούσατε να κάνετε για να βελτιωθεί το σημερινό σύστημα. Επανέρχομαι στην ερώτηση που έκανε ο Χιόκμαρκ στην ΙΚΕΑ, αλλά αφορά και τους δυο σας. Εμείς είμαστε 28 χώρες στην Ένωση με 28 διαφορετικούς εταιρικούς φόρους. Κανονικά, εάν το αντικαταστήσουμε από ένα και μοναδικό σύστημα, είναι καταπληκτική, τρομακτική απλοποίηση. Ρωτήσαμε και άλλες πολυεθνικές εταιρείες. Ήταν πάρα πολύ ε, υπέρμαχες. Έχω την αίσθηση ότι το σύστημα του franchise σας επιτρέπει να ζείτε πιο εύκολα από ότι κάποιοι άλλοι. Δεν είναι καθόλου κριτική αυτό, ούτε φιλοφρόνηση. Είναι μια τεχνική ερώτηση. Σας βοηθάει περισσότερο, σας απλουστεύει τη ζωή αυτό από άλλα συστήματα με τα 28 διαφορετικά φορολογικά συστήματα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι προφανές ε, πως πιστεύω ότι αυτή η απλούστευση θα ευνοήσει τις επιχειρήσεις και σίγουρα θα προκύψει. Γιατί είναι πολύ εύκολο το να προσπαθήσει και να καταλάβει και να προσπαθήσει κάποιο να συμμορφωθεί με ένα σετ κανόνων και όχι 28 διαφορετικά. Σε σχέση με αυτά που ακούσαμε νωρίτερα και από απάντηση τη κυρία Κοντζόναλτ, ούτε εμεί έχουμε τον καταμερισμό για το σύνολο των ΦΠΑ, των φόρων επί των μισθών κτλ. διότι δεν ε, τους πληρώνουμε ε, αυτούς τους φόρους ουσιαστικά. Όπως σας είπα, όμως, όταν μιλάμε για την ανάπτυξη, για τις δραστηριότητες αναπτυξιακές, ε, συμβάλλουμε έτσι στους φόρους, γιατί δημιουργείται ΦΠΑ, γιατί καταβάλουμε τους μισθούς για... τους φόρους για τους μισθούς και το ίδιο ισχύει και για τους προμηθευτές μας, τους δίνουμε δουλειά. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι δεν μπορεί να θεωρηθεί αυτό ως εισόδημα. Υπερβάωσε, είναι ανυπόμονη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Προς την κυρία Μιέτς ε, θα ήθελα να υποβάλω την ερώτηση, αλλά την ίδια θα μπορούσα να υποβάλω και στην ΙΚΕΑ. Τέσσερις είναι οι ερωτήσεις. Πρώτον, για να επανέλθω ε, στην ε, μετανάστευσή σας, ε, το διπορικό μέσο Ελβετίας. Αλλά ε, φεύγει η κυρία από το Μακδόναλτς, τι να την κάνω την ερώτηση, δεν με ακούει. Yes, but I'm asking the question to McDonald's. Okay. I said I could also raise the question. Ε, έλεγα θα μπορούσα ε, να, ε, το, να υποβάλω την ερώτηση και στην οικία, αλλά προτιμώ στο McDonald's. Ε, θα, το πω, θα τα πω στα γαλλικά, καλύτερα για αυτούς που με ψηφίζουν και ενδιαφέρονται για αυτό το ζήτημα. Λοιπόν, γιατί πρέπει να περάσετε από την Ελβετία. Καταλαβαίνω ότι πληρώνετε του φόρους στο Λουξεμβούργο, αλλά γιατί πριν πάτε ΣΥΠΑ πρέπει να περάσετε από την Ελβετία. Και όταν πάτε εκεί, με πώς ε, προσγειώνεστε στο Delaware, από ποιου και τι σημαίνει αυτό που είπατε για την Ελβετία, δηλαδή Εάν εμεί θεωρήσουμε ότι πρέπει να περάσετε από άλλη χώρα, δεν θα έχετε πρόβλημα. Γιατί η Ελβετία, γιατί συγκεκριμένα η Ελβετία. Δεύτερον, μπορείτε να μας πείτε για το reporting, country reporting, δηλαδή την υποβολή εκθέσεων αναχώρα. Γιατί έχετε τόσες ε, ε, επιφυλάξεις και ενστάσεις σε σχέση με την πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπής ως προς το δημόσιο χαρακτήρα αυτών των εκθέσεων ε, ε, γιατί υπάρχουν και άλλοι τομείς ε, όπως ε, ο τραπεζικός τομέας διότι πιστεύουμε ότι αυτές οι επιχειρήσεις δεν θα μπορούσαν να, να λειτουργήσουν διαφανέστερα και όταν μας λέτε ότι Ε, ότι υπάρχουν επιχειρήσεις που κάνουν λόμπινγκ για να ισχύσει ένα άλλο σύστημα πέρα από αυτό του Σε θα μας ενδιαφέρει να μα το πείτε. Δεύτερον, για το εφαρμοστέο σύστημα. Κυρία Γέιτς, είπατε ε, θέστε στους κανόνες και εμείς θα τους εφαρμόσουμε στην Ευρώπη αλλά και αλλού στον κόσμο εμείς ε, ανησυχούμε διότι φοροδιαφεύγεται. Αν σας έλεγα λοιπόν ότι Αύριο θα είναι εφαρμοστεί το γαλλικό δίκαιο. Τι θα λέγατε λοιπόν. Ποια θα ήταν η απάντησή σας. Δηλαδή θα ήταν ένα, μία δέσμη κανόνων, ε, αλλά θα ίσχυε το γαλλικό δίκαιο. Πώς θα αντιδρούσατε. Και τελευταία ερώτηση, μας είπε ότι πληρώνετε πολλούς φόρους. Τι γίνεται όμως όταν αφαιρείτε το ΦΠΑ. Εμάς μας ενδιαφέρει ο φόρος για τις επιχειρήσεις, όχι το συνολικό ποσό. Έχετε το λόγο για να απαντήσετε, κυρία μου. Δεν είμαι σίγουρη ότι κατάλαβα την ε, τελευταία ερώτηση, αλλά όσα κατάλαβα, όσα κατάλαβα θα απαντήσω, εν Για τις εκθέσεις αναχώρα, για, δεν έχουμε προτίμηση για την εμπιστευτικότητα ή τη δημοσίευση. Εμείς θα εφαρμόσουμε τους κανόνες όπως και σήμερα. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να συμμορφωθούμε με τους κανόνες. Για την Ελβετία και τη ΣΥΠΑ. Ε, είναι η δομή αυτή που έχουμε για τις άδειες. Έχουμε μια, ένα λειτουργικό ε, υποκατάστημα στην ε, επιχειρησιακό υποκατάστημα στην Ελβετία και εκεί ασχολούνται με την στρατηγική κατευθύνσης γραμμές για την καινοτομία και για την ε, πολιτική που εφαρμόζουμε γενικότερα. Η Ελβετία δεν εισπράττει ρόγελ Γι' αυτό το σημείο πριν έρθει σε Περβάος, αποφασίσαμε ότι θα μας στείλει μια γραπτή ερώτηση γι' αυτό το... Ε, γραπτή απάντηση, συγγνώμη. Ε, αυτό θα κάνω ακριβώς. Και γιατί έχετε δώσει τόσους ενδιασμούς και ενστάσεις ε, για την πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπής, ήταν η δεύτερη ερώτηση. Μα και ακόμη και για την κοινή ενοποιημένη βάση θα εφαρμόσουμε την ομοθεσία. Θέλουμε να έχουμε τη βέλτιστη δυνατή απάντηση. Τώρα είναι περασμένη η ώρα και έχουμε μιλήσει για συνθήκες ανταγωνισμού, δεν χρειάζεται να τα ξαναλέω. Πρόεδρος, μπορείτε για το συνολικό φόρο να μας πείτε πώς επιμερίζεται ΦΠΑ, εταιρικός φόρος κτλ. Δηλαδή τάξη μεγέθος, όχι πόσο. Δεν τις έχω τις πληροφορίες εδώ. Με σοκάρετε, λέει η κυρία Περές, διότι λέτε πληρώνουμε πάρα πολλούς φόρους στην Ευρώπη και δεν ξέρετε πόσα είναι ΦΠΑ και πόσα είναι CCTB. Τώρα πλάκα κάνετε. Μα συγγνώμη, ο φόρος ε, καταβάλλεται από τους πελάτες μας ο ΦΠΑ και μετά ε, το είπε ο συνάδελφος δεν είναι υποχρέωση της εταιρείας ε, να δίνει αυτά τα στοιχεία. Εγώ μπορώ να σας πω ότι πληρώνει η McDonald's Corporation και δεν θα επανέλθω, πληρώνουμε πολλούς φόρους. ΦΠΑ. Όταν, ε, όταν είναι επιτυχημένες οι δραστηριότητες μας στην Ευρώπη, τότε πληρώνουμε και περισσότερο ΦΠΑ. Δεν τα έχω όμως τα νούμερα. Θα μας τα στείλετε γραπτός. Θα δω αν μπορώ να τα βρω. Λοιπόν, από τους συντηρητικούς και μεταρρυθμιστές, ο κύριος Κρασνοτεύσκη. Ευχαριστώ πολύ. Αν μου επιτρέπετε θα μιλήσω πολωνικά εγώ για αλλαγή. Ευχαριστώ. Πρέπει να σας πω ότι με εντυπωσιάζει πραγματικά η ευημερία όλων των εταιριών που ακούσαμε και η παρουσία όλων των εκπροσώπων με έχουν εντυπωσιάσει αυτά που δηλώνετε ότι θα τηρήσετε τους νέους νόμους όποιοι και να είναι αυτοί. Έχω μια ερώτηση. Οι εταιρείε σας δεν μπορεί να αγνοούν ε, την αυξανόμενη κοινωνική διαμαρτυρία και τη δυσφορία του κόσμου ε, στις κοινωνίες μας, στις κυβερνήσεις μας υπάρχει ένας άλλος που επικρατεί ε, και σε σχέση με τα όσα λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ερωτώ, τι δράσεις εσείς αναλαμβάνετε στην εταιρεία σας, ο καθένας, για να ανταποκριθεί σε όλες αυτές τις νέες ανάγκες και τα νέα δεδομένα. Ο κόσμος έχει αγανακτήσει, έχει απειβδίσει. Θα έχετε συζητήσει αυτά. Ε, μιλήσατε για απλούστευση, για διαφάνεια, όλα αυτά μας τα είπατε, αλλά ε, πολύ συγκεκριμένα τι σημαίνουν αυτά. Και ε, παίρνετε και εσείς τέτοια βήματα, κάνετε τέτοια βήματα μάλλον πριν να αποφασίσουμε εμείς πριν νομοθετήσουμε σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτά. Ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος, ο κύριος Χάνσεν. Θέλετε να αρχίσετε εσείς αυτή τη φορά. Yes, uh, as, I... Όπως είπα και στην αρχική μου τοποθέτηση, καλά και εμείς τυφλοί δεν είμαστε, ούτε κοφοί. Βλέπουμε τις συζητήσεις που γίνονται και τις ακούμε και στην κοινωνία και στο κοινοβούλιο σας. Και γι' αυτό ενδιαφερόμαστε πάρα πολύ ε, έτσι ώστε από κοινού να βρούμε μια κοινή και ε, καλή λύση για το μέλλον. Κυρίως αυτό που μας ενδιαφέρει είναι απλότητα και η σαφήνεια. Για να μην μπορούν να τα καταλάβουν όσοι έχουν διδακτορικό μόνο, είμαστε και εμείς σε θέση να καταλαβαίνουμε τους νόμους και να τους στηρούμε, να συμμορφωνόμαστε. Αυτό μας ενδιαφέρει να συμβεί. Και όπως είπα στην αρχή, όλοι βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποιοι νομοθέτες που παίρνουν αυτές τις αποφάσεις και εμείς και άλλοι στην κοινωνία μας τους εφαρμόζουμε. Τυφλοί πάντως δεν είμαστε ούτε κοφοί. Βλέπουμε και εμείς τι συμβαίνει. You see, my Εγώ άλλο πράγμα ρώτησα. Δεν λέω τι κάνετε εσείς και ποιος είναι ο νέος κανονισμός. Είναι πολύ περίπλοκο αυτό, πώς να το πω για έναν άνθρωπο μέσης νοημοσύνης να καταλάβει πώς διαρθρώνεται μια τέτοια εταιρεία. Εγώ σας ερωτώ, εσείς τι κάνετε για μας, για να μπορέσουμε εμείς να καταλάβουμε πώς πληρώνετε φόρους, πώς το οργανώνετε όλο αυτό, όλη αυτή την πίσνα, διότι είναι και τη ζούγκλα αν ρίξει κανείς μια ματιά για να καταλάβει τι γίνεται. Πελαγώνει, είναι ολόκληρα δίκτυα και πλοκάμια και σας ρωτώ εσάς τους δύο τι κάνουν οι δικές σας εταιρείε για να μας πείσετε εμάς τους βουλευτές δηλαδή, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά και την κοινή γνώμη ότι έχετε σαφή ειλικρινή δομή. Και ορίστε, σας δείχνουμε για να ε, καταλάβετε και με τρόπο εύληπτο ο καθένας και κάθε μια από τους ψηφοφόρους μας να καταλαβαίνουν ότι πληρώνετε τους φόρους σας όπως και μια νομοταγής μικρή εταιρεία. Μπορείτε να απαντήσετε, θέλετε να απαντήσετε, μπορώ, ναι, ναι. Και χαίρομαι για την ερώτηση, γιατί έχει να κάνει με την απλούστευση που μας ε, ενδιαφέρει και επίσης εκτιμώ το γεγονός ότι Κατανοώ μάλλον αυτό που λέτε ότι τα συστήματα franchising μπορεί να είναι περίπλοκα. Προσπάθησα να σας εξηγήσω όσο μπορούσα πιο απλά ότι είναι ένα σύστημα που έχει κάποιος ε, ένα σήμα που λέγεται IKEA και υπάρχουν πολλοί που νοικιάζουν αυτό το σήμα παγκοσμίω. Είναι απλό το μοντέλο γιατί πρέπει να συνεργαζόμαστε για να προχωρούμε και να είναι αμοιβαία επωφελής αυτή η κατάσταση και για εκείνον που εχωρεί το δικαίωμα και για εκείνον που το χρησιμοποιεί. Μπορεί να είναι δύσκολες οι λέξεις στα αγγλικά, αλλά δεν είναι δύσκολες οι έννοιες. Προσπάθησα να το εξηγήσω και ελπίζω να τα κατάφερα. Παρακαλώ, κυρία μου. Συμφωνώ με πολλά από αυτά που υπόθηκαν. Χαίρομαι ιδιαίτερος που ε, βρίσκομαι μεταξύ σας για δεύτερη φορά ε, και προσπαθώ να δώσω περισσότερες πληροφορίες προς τα έξω ε, σχετικά με το τι κάνουμε. Θεωρούμε ότι πολλά στοιχεία είναι θετικά στην εταιρεία μας. 25% της δραστηριότητές μας αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για 8.000 καταστήματα τα οποία δίνουν δουλειά σε πολίτες, άνδρες και γυναίκες. Η πολιτική μας απέναντι στους franchisees είναι συγκεκριμένη. Τους δίνει πρόσβαση ε, σε όλες τις αναβαθμίσεις γνώσεων, κατάρτισης, ε, ιδιοκτησίας. Ε, εμείς μοιραζόμαστε μαζί τους την άποψη σχετικά με το φαγητό, σχετικά με τις διατροφικές συνήθειες, σχετικά με ένα σωρό πράγματα. Στην ουσία αυτό που κάνουμε είναι πολύ συγκεκριμένο και βεβαίως ε, ε, δεν έχουμε κανένα λόγο να μην συζητήσουμε μαζί σας και για ενδεχόμενες απώλειες. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να είναι ίσες ε, οι συνθήκες και ισότιμες οι συνθήκες και να αφορούν όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων. Ευχαριστώ πολύ. Μία τελευταία ερώτηση από πλευράς του κυρίου Ντεμάζη που είχε θέσει υποβάλει ένα συγκεκριμένο ερώτημα το οποίο όμως δεν απαντήσατε. Ε, είχαμε τη χαρά να σας ε, ε, έχουμε μαζί μας πριν μερικούς μήνες στη διάρκεια της πρώτης ακρόασης. Δεν είχατε αναφέρει το γεγονός ότι είχατε κάνει μια συμφωνία ruling με το Λουξεμβούργο. Γιατί τότε δεν αναφέρθηκε το θέμα. Αυτή είναι η ερώτηση του κυρίου Ντεμάζη δεν είμαι σίγουρη ότι ρωτήθηκα για το, για το κατά πόσον υπήρξε ruling με το Λουξεμβούργο. Κοιτάξτε, αυτά τα θέματα ελέγχονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επομένω δεν μπορώ να τα συζητήσω. Όσον αφορά νέε συμφωνίε, new business arrangements ή όσον αφορά ε, τέτοια παρόμοια πράγματα, το σημαντικό είναι να υπάρχει σαφήνεια. Ναι, εντάξει, ξέρουμε τι είναι το ruling, λέει ο πρόεδρο. Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο μορφέ όμω. Ε, υπάρχει ε, μία μορφή η οποία αναφέρεται στις κρατικές επιδοτήσεις και μία ε, τύπου ε, αυτών που υπέγραψε η McDonald's. Δεν ρωτάω αυτό λέει ο Πρόεδρος. Υπήρξε συμφωνία ruling ανάμεσα στο Λουξεμβούργο και το ε, ε, και το, την McDonald's και εσείς δεν μας το αναφέρατε. Ναι, ε, απάντηση, νομίζω ότι δεν ερωτήθη, γι' αυτό δεν απήντησα. Πολύ ωραία, ολοκληρώσαμε και το δεύτερο πάνελ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συμμετέχοντες στα δύο πάνελ. Το μήνυμα για τους καλεσμένους μας, το καταλάβατε νομίζω, είναι ότι εμείς αλλάζουμε εποχή. Και το τελευταίο ερώτημα του κυρίου Κρασδεύσκη ήταν στην ουσία μία έκκληση, δεν ήταν επίκριση, δεν ήταν κριτική, εάν κατάλαβα καλά και όλα αυτά που θέλατε να πείτε, ήταν μία έκκληση στην ουσία. Ε, καταλαβαίνετε ότι πλέον μετά τα σκάνδαλα τα οποία έλαβαν χώρα, μετά από την ε, ε, οικονομική κρίση, μετά από το ξέσπασμα ε, των, των ε, συμπολιτών μας, τον θυμό τους απέναντι στον τρόπο λειτουργίας των μεγάλων επιχειρήσεων, τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονται οι πλούσιοι με την ευρύτερη έννοια του χώρου. Καταλαβαίνετε λέω ότι μετά από όλα αυτά κάποιοι νόμοι, κάποιες πρακτικές που λειτουργήσαν τα 20 τελευταία χρόνια δεν γίνονται πλέον ανοιχτοί από τους πολίτες. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι εμείς, εμείς που ε, κάνουμε τους νόμους θα πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και πρέπει να πω ότι η δικιά σας ευθύνη, για να μην πω το, το δικό σας συμφέρον είναι να αλλάξετε κι εσείς πρακτικές. Πριν από κάποιες δεκαετίες ε, ε, εισάγατε στην πολιτική των ομίλων σας την έννοια της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης Έχετε λοιπόν αναλάβει και έχετε αναγνωρίσει ότι έχετε κάποιες υποχρεώσεις απέναντι στους μισθωτούς σας όσον αφορά τις εργασιακές συνθήκες, τη συμμετοχή στο κεφάλαιο, τις αμοιβέ τους, τις συνθήκες υγιεινής τη συμμετοχή στην διαδικασία λήψης απόφασεων κτλ. Πιο πρόσφατα κατανοήσατε ότι σαν ε, ε, σαν εταιρείε ε, παρούσες σε ολόκληρο τον κόσμο ότι έπρεπε να ενδιαφερθείτε και για το περιβάλλον. Ανακύκλωση, κυκλική οικονομία, προστασία της βιοπικιλότητας, επαναχρησιμοποίηση, μείωση απορριμμάτων και αποβλήτων και τα λοιπά και όντως ε, αυτό το κάνατε σημαία στις ε, επιχειρήσεις σας ε, και για το, για το McDonald's η ποιότητα των πρώτων υλών και για το IKEA προστασία του περιβάλλοντος, πράσινη συνείδηση και τα λοιπά είναι σημαίες για σας. Αυτά τα μετατρέψατε λοιπόν σε επιχειρηματικά σύμβολα Νομίζω ότι προς το συμφέρον σας είναι πλέον να πείτε και να έχετε το δικαίωμα και τη δυνατότητα να πείτε ότι είμαστε ε, ε, συνειδητοποιημένοι ε, υποδειγματικοί φορολογούμενοι. Ε, στην ε, παρούσα ε, παγκόσμια συνθήκη όντως τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα έτσι ώστε να κατανοήσουμε αυτούς τους μυστικούς δρόμους της φορολογίας ανάμεσα από εταιρείες θηγατρικές, δευτερεύουσες έδρες κτλ. Αλλά, αλλά νομίζω ότι πλέον είναι σαφές ότι και στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και βάσει της BEPS σε παγκόσμιο επίπεδο ε, ε, πρέπει λέω να γίνουν κάποιες μεταρρυθμίσεις και είναι προς το συμφέρον το δικό μας αλλά και προς το δικό σας γιατί προφανώς είναι προς το δικό σας συμφέρον να ε, υπάρχει μια βάση η οποία θα είναι παρόμοια σε παγκόσμιο επίπεδο και φυσικά δεν μας ενδιαφέρει εμάς εδώ να σας βάζουμε συνέχεια δυσκολίες βάζοντας συγκεκριμένους κανόνες εάν στα άλλα μέρη του κόσμου της υφηλίου ε, δεν ακολουθούνται και δεν επιβάλλονται οι ίδιοι ε, κανόνες. Αυτό που είναι σημαντικό να καταλάβουμε όλοι είναι ότι αλλάζουμε εποχή. Θα δώσω τώρα το λόγο ε, στον εισηγητή μας για να βγάλει τα τελικά συμπεράσματα. Θα ήθελα και εγώ από τη δικιά μου μεριά να ευχαριστήσω τους εκπροσώπους των ε, εταιριών ε, που ήταν μαζί μας, την Google, την Apple, ε, την IKEA και τη McDonald's. Είναι ενδιαφέρον γιατί ακούσαμε πολλές φορές να, αναφέρεται, ε, να αναφέρονται κάποια πράγματα. Ε, δηλαδή μας είπε η Google ότι χρησιμοποιεί κάποιες ε, φορολογικές πρακτικές οι οποίες είναι γνωστό, γνωστές σε όλο τον κόσμο. Είτε αυτές λέγονται double iris, είτε λέγονται Ολλανδικό sandwich, είτε οτιδήποτε. Δηλαδή ότι υπάρχουν αυτές οι δυνατότητες τις οποίες χρησιμοποιούν οι μεγάλες εταιρείες. Επομένως, από τη στιγμή που εσείς ζητάτε ε, σαφήνεια και ε, ε, διαφάνεια των νομοθετημάτων και εμείς σας ζητούμε το ίδιο. Θέλουμε να υπάρχει σαφήνεια, θέλουμε να υπάρχει διαφάνεια και έτσι ώστε το κέρδος, τα κέρδη να φορολογούνται εκεί που παράγονται. Αυτή είναι η πρώτη μου ε, παρατήρηση. Βεβαίως η βάση ως ΑΜΠΕΠΣ είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό αλλά δεν έχει έννοια εάν δεν γίνονται οι εκθέσεις αναχώρα ε, γιατί αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να είναι ένα σύστημα, αντα... ένα σύστημα το οποίο θα βασίζεται στην ανταλλαγή των πληροφοριών όπως άλλωστε και τα συστήματα της ενιαίας φορολογικής βάσης, το CCTB. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση, αλλά πρέπει να σας πω ότι η νομοθεσία ε, ε, του ανταγωνισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και γενικότερα ε, καλύπτει, ε, καλύπτει τις ε, την εταιρική φορολογία και είναι πάρα πολύ σημαντικό σε αυτά τα πλαίσια να μην υπάρξει καμία στρέβλωση του ανταγωνισμού. Όπως είπα και στην αρχική μου παρέμβαση, είναι γεγονός ότι οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις πληρώνουν τουλάχιστον 13% επιπλέον φορολογικό βάρος ε, ε, από ότι, οι μεγάλες ε, εταιρείες οι οποίες έχουν την δυνατότητα να προσφύγουν σε διάφορα τεχνάσματα. Εγώ λοιπόν σας ζητώ να μην εμποδίσετε την απλούστευση της νομοθεσίας, να μην εμποδίσετε την μεγαλύτερη σαφήνεια όταν θα έρθει η συζήτηση στον όσα. Παρακαλώ πολύ να διευκολύνετε αντιθέτως την κατάσταση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σιγητά. Θα παραμείνουμε σε επαφή. Θυμίζω ότι περιμένουμε γραπτές ε, απαντήσεις από την ΙΚΕΑ αφενός για την υποτιθέμενη έκθεση των υποτιθέμενων ε, πρασίνων του πρασίνου που υποτίθεται ότι δεν είναι παρόν πια και από εσά, κυρία μου σε ό,τι αφορά ε, την ασφαλιστική δραστηριότητα στις Βερμούδες. Κάποιοι συνάδελφοι δεν γνωρίζουν ότι οι Βερμούδες που έχουν μια φήμη ε, αρκετά εκρηκτική από πλευράς ε, φορολογικής είναι ένα κέντρο ασφαλιστικό, ιδιαίτερα για τις Ηνωμένε Πολιτείε. Να μας διευκρινίσετε λοιπόν τι ισχύει για το δικό σας όμιλο ε, και μας τάξατε και μια απάντηση για τα ταξίδια που κάνουν διάφορα ποσά από την Ελβετία στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω Delaware. Μπορεί να μας το στείλετε και σε σκίτσο αυτό. Δεν υπάρχει άλλο θέμα στη μέση διάταξη. Λοιπόν, ραντεβού για τα μέλη της Επιτροπής μας και όλους όσοι ενδιαφέρονται για τις εργασίες μας. Στις 21 Μαρτίου το απόγευμα θα δούμε τι ώρα αναλόγως με το πόσες ακροάσεις θα έχουμε. Και θα ε, αφιερωθούμε στις τράπεζες, σε λήξη συνεδρίες.